Welcome Καλώς ορίσατε όλοι. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω μετά τις διακοπές. Σας είδα βέβαια και στην Ολομέλεια. Αλλά είναι μεγάλη μου τιμή επίσης που είναι εδώ μπροστά μας και ο Υπουργός Αθλητισμού του Λουξεμβούργου ο κύριος Ρόμαν Σνάιντερ. Δεν είναι μόνο αθλητισμού, αλλά και κοινωνικής κοινωνικών ασφαλίσεων και ανάπτυξης. Ε, ε, τα υπόλοιπα θα τα πω ιταλικά, αλλά τα πρώτα δύο σημεία να έτσι. Τώρα τα πρώτα δύο. Ε, μετά ο υπουργό. Και τώρα λοιπόν πρώτα πρώτα ελπίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη το πρώτο, το πρώτο σημείο και το πάμε στο δεύτερο ήταν στο τρίτο έγκριση των πρακτικών έχουμε κάποιες ε, παρατηρήσεις αλλιώς ε, προχωρούμε οπότε θα δει απλώς να σας αναφέρω ότι σήμερα έχουμε σε γαλλικά, ιταλικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, διερμηνία ε, τσεχικά, εστονικά, ουγγρικά, ε, πολωνικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Η συνεδρίαση μας δεν πρόκειται να μεταδοθεί στο ίντερνετ. Πριν προχωρήσουμε χθες αμέσως στα, στα της ε, συνάντησης με τις προτεραιότητες του Υπουργού για τον Αθλητισμό, είναι σήμερα η πρώτη μας συνεδρίαση με τις διακοπές. Οπότε πρέπει να σας αναφέρω ότι αυτό το δίμηνο το οποίο πέρασε το λέγαμε με την κυρία Μπόκοβα και θέλαμε ακριβώς να διατυπώσουμε τον προβληματισμό μας για τα όσα γίνονται κοντά μας εδώ στην Συρία είχαμε την ανθρωποκτονία ενός εξαιρετικού αρχαιολόγου προσπάθησε να την Παλμύρα και την εκεί πολιτιστική κληρονομιά κύριος Καλέντα Λάσσα. Οπότε νομίζω ότι και εμείς θα πρέπει όπως ε, και άλλοι να τον σκεφτούμε. Και έχουμε επίσης μια συνάντηση που έχει οργανώσει η Λουξεμβουργική Προεδρία που θίγει και αυτό το ζήτημα. Τώρα επομένω θα σα τον Υπουργό κύριο Σνάιντερ. Σα αναφέρω ότι πρώτα πρώτα τον καλωσορίζουμε. Μιλήσουμε για τι προτεραιότητε τη Προεδρία σα. Προτεραιότητε που ταυτίζονται με ό,τι απασχολεί εμάς και κάναμε ένα εργαστήριο πρόσφατα με κάποιους ειδικού. και θα γίνει επίση άλλο πρόκειται να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες οπότε και θα μας πείτε τι βλέπετε όσον αφορά το πώς θα υπάρχει ευρύτερη συμμετοχή στον αθλητισμό από όλες τις ηλικίε. Και έτσι θα αναπτύσσονται οι ικανότητες όλων στον αθλητισμό. Και πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο βέβαια και απαιτεί την σωστή διακυβέρνηση. Ξέρω ότι εσείς ε, ασχολείστε πάρα πολύ με την καταπολέμηση του ντόπινγκ και εμεί σαν Επιτροπή Πολιτισμού έχουμε ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα και είχαμε την έκθεση φύσας για τον αθλητισμό. Εκεί καλύψαμε τις αρμοδιότητες που έχουμε για τον αθλητισμό στην Ευρώπη δυνάμεις συνήθως της Λισαβόνας. Και επίσης μέσω του Έρασμου ΣΥΝ έχουμε ένα ολόκληρο πρόγραμμα του υπηρεσίου του αθλητισμού μέχρι το 2020. Θα μιλήσουμε και για την ε, εβδομάδα του αθλητισμού, την ευρωπαϊκή. και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα, να προβάλλουμε καλύτερα την ευρωπαϊκή πολιτική αθλητισμού και το πώς θα έχουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο αθλητισμού. Και είπαμε για το ε, εργαστήριο το οποίο είχαμε όσον αφορά τον αθλητισμό, οπότε έρχεται αυτό που θα μας αναπτύξετε να ε, κολλήσει σε αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Έχετε τώρα το λόγο κύριε Υπουργέ. Euh, euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτέ. Πολύ σημαντικό σημείο μέρος της Προεδρίας μας είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα μεταξύ των υπολείπων προτεραιοτήτων μας. Γι' αυτό θέλησα να κάνουμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ καταρχάς που με καλέσατε για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητές μας στον τομέα του αθλητισμού για το εξάμεινο αυτό. Για μένα δεν είναι απλή τυπικότητα, αλλά όπως σας είπα και πριν θέλω να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο με την Επιτροπή σας που παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των θέσεων του Κοινοβουλίου για τον αθλητισμό. Υπάρχει λοιπόν διαθεσμικός διάλογος και αυτό είναι σημαντικό προς το συμφέρον βέβαια κυρίως του πολίτη. Και η Λουξεμβουργική Προεδρία θέλει αυτό να είναι το κέντρο βάρος κάθε πολιτικής. Στον τομέα του αθλητισμού αυτά μεταφράζονται στη θέληση να καλύψουμε μία πτυχή ακόμη άγνωστη του θέματος, δηλαδή την προώθηση των σωματικών δραστηριοτήτων στους μικρούς παιδες μέχρι και κάτω των τριών ετών για να μην έχουν στη συνέχεια της ζωής τους καθιστική ζωή. Από αυτό θα αρχίσουμε λοιπόν και θα δούμε μετά ποιες είναι οι υπόλοιπες προτεραιότητες. Αρχίζουμε πάντως με την προώθηση των σωματικών δραστηριοτήτων και της κίνησης των παιδών. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει πει ότι η σωματική άσκηση είναι ε, πολύ σημαντικός παράγοντας για την καταπολέμηση της, των πρώιμων θανάτων και πολύ αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης της παχυσαρκίας. Ακόμη και όλο και περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ ψυχικής υγείας και σωματικής δραστηριότητας. Επίσης ξέρετε ότι η φυσική δραστηριότητα δεν έχει πτώσει μόνο επί της υγείας ε, των ατόμων αλλά και ολόκληρων των συστημάτων υγείας των χωρών. Το ξέρω και ως υπουργό. Υπολογίζουμε ότι περίπου 7% των προϋπολογισμών υγείας των χωρών μελών αφορούν ασθένειες σχετικές με την παχυσαρκία γιατί η καθιστική ζωή έχει αρνητικές συνέπειες και δεν αφορά αυτό μόνο τους ενήλικες ούτε απομονώνουμε μόνο το θέμα της παχυσαρκίας. Υπάρχουν και τα μειοσκελετικά προβλήματα στην Ευρώπη, ακόμη και στα νέα παιδιά. Και οι αριθμοί δείχνουν ότι στις βιομηχανικές χώρες και παιδιά κάτω των 5 ετών έχουν, ε, εμφανίζουν φαινόμενα παχυσαρκίας και υπερβολικού βάρους. Μέχρι και 12% το 2010 και ίσως φτάσει αυτό το ποσοστό το 15% το 20%. Το Λουξεμβούργο βρίσκεται σε περίπου 10% παιδιών με τέτοια προβλήματα. Επομένως προτεραιότητα της Προεδρίας είναι ότι οι φυσικές δραστηριότητες δεν είναι μόνο θέμα υγείας αλλά αποφυγής ασθενειών αλλά και ανάπτυξη της μυϊκής δύναμης, τη συντονισμού των μειών και της ψυχικής υγείας καθώς και της ε, ισορροπίας του οργανισμού γενικότερα. Μελέτες δείχνουν σαφώς ότι τα παιδιά αρχίζουν να αθλούνται, που αρχίζουν να αθλούνται από μικρά έχουν καλύτερα σχολικά αποτελέσματα και καλύτερη συμπεριφορά διαγωγή. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τον το ρόλο που έπαιξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πρωτοπόρος από το 2007 για το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία και μετά στο ψήφισμα ένωνυμ τόνιζε ήδη ότι πρέπει να δοθεί σημασία στον αθλητισμό για τα παιδιά μικρής ηλικίας για να μπορέσουν να αρχίσουν όσο δυνατόν νωρίτερα να ασχολούνται με κάποια φυσική δραστηριότητα. Η προώθηση λοιπόν των δραστηριοτήτων αυτών είναι κάτι που, με το οποίο ασχολούνται πολλοί στην Ευρώπη και στο οποίο δίνουμε όλο και περισσότερη σημασία ακόμη και από το Συμβούλιο γιατί το ενδιαφέρον για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που αθλούνται είναι πολύ μεγάλο. Θελήσαμε λοιπόν κατά τη Λουξεμβουργική Προεδρία να επιμείνουμε στη σημασία που έχει να αποκτήσει κανείς από τη γέννηση του ήδη έναν ενεργό τρόπο ζωής και στο Συμβούλιο του Νοεμβρίου θα καταθέσουμε σχετικές προτάσεις ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα σχολεία και οι αρχές των χωρών μελών για τη σημασία του αθλητισμού. Τα συμπεράσματα θα καταλήξουν και σε συστάσεις εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου που κατατέθηκαν ήδη από τον Ιούνιο. Είναι καινούριο τρόπος αυτός σύλληψης των πραγμάτων Σήμερα λέμε στα παιδιά μην κουνιέσαι. Στο μέλλον θα λέμε κουνήσου, κουνήσου. Δεύτερο θέμα. Πολύ σημαντικό επίσης για την Προεδρία μας, κυρία Πρόεδρε, είναι η εκπροσώπηση και ο συντονισμός της Ένωσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Καταπολέμησης του του ντοπάζ. Πρόσφατα αποδείχτηκε ότι το φαινόμενο αυτό δεν βλάπτει μόνο τους ίδιους τους αθλητές αλλά και την εικόνα του αθλητισμού την ίδια. Και γι' αυτό θέλουμε η Ευρώπη να ακουστεί με δυνατή φωνή. Το τωρινό σύστημα εκπροσώπησης και συντονισμού στην Ένωση από την οργάνωση αυτή βασίζεται στις συστάσεις του Συμβουλίου του 11 που πρέπει να ενημερωθούν το 15. Με μεγάλη χαρά λοιπόν πρότεινα να γίνει η ενημέρωση αυτή κατά τη Λουξεμβουργική Προεδρία πόσο μάλλον που για λίγους ακόμη μήνες θα προεδρεύουμε ως προεδρία και στην οργάνωση αυτή έτσι ώστε οι ευχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ληφθούν περισσότερο υπόψη εκεί. Κάναμε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Υπουργών Αθλητισμού σε άτυπη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις αρχές του Ιουλίου. Δεν διαγράφηκε βέβαια καμία συνένεση για την αλλαγή της εκπροσώπησης, αλλά πολλοί συνάδελφοι μας ζήτησαν να βελτιώσουμε το συντονισμό στην Ευρώπη ενώπιον των εθνικών αρχών καταπολέμησης του ντόπινγκ. Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες. Η Λουξεμβουργική Προεδρία καλεί τακτικά τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη εγκρίνει έναν εθνικό κώδικα αντιντόπινγκ να το πράξουν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Επίσης τον Νοέμβριο θα κατατεθούν οι προτάσεις της Ένωσης για την οργάνωση αυτή. Ο Βέλγος συνάδελφός μου Φίλιπ Μόιτενς ε, λύγει λίγη η θητεία του στην Προεδρία του οργανισμού αυτού και πρέπει να εκλεγεί ένας νέος εκπρόσωπος εκ μέρους της Ευρώπης για να παραμείνει δυνατή η φωνή της. Τρίτο σημείο των προτεραιοτήτων μας. Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης για μας. Η διπλή καριέρα για τους αθλητάς ώστε να μπορούν να συμφιλιώνουν τον αθλητισμό τους υψηλού επίπεδου με την εκπαίδευσή τους, ανώτερη ή ανώτατη. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν μέτρα, αλλά θεωρούμε ότι παραμένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Η ευρωπαϊκή ιδίως να γινουν η ευρωπαικη ιδίω διασταση του προβλήματος αυτού, διότι σήμερα οι αθλητές έχουν μεγάλη κινητικότητα για να συμμετέχουν στους διάφορους αγώνες με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες άσκησης. Άρα για να μπορέσει να, κανείς να προπονηθεί μένοντας πολύ καιρό στο εξωτερικό πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να συνεχίσει και τις σπουδές του. Άρα η Προεδρία θα εξετάσει αυτό το θέμα σε μια πρώτη άτυπη συνεδρίαση ανταλλαγή απόψεων αύριο και μεθαύριο στο Λουξεμβούργο με διευθυντές αθλητικών προγραμμάτων και μετά μια πρόσθετη διάσκεψη την οποία θέλω και να σας καλέσω είναι ενδιαφέρουσα με υψηλού επίπεδου αθλητάς ευρωπαϊκής σημασίας. Ας μην επεκταθώ τώρα σε αυτή τη διάσκεψη των, την άτυπη των δύο επομένων ημερών αλλά θα αναφέρω ότι η Προεδρία θέλει να συζητήσει και ένα θέμα ανταλλαγής βελτίστων πρακτικών ανεξαρτήτως θρησκείας, πολιτισμού και λοιπά και μεταναστευτικών αρχών οι προελεύσεων. Θα ήθελα επίσης να σας δηλώσω ότι θέλουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις που έχουμε ως δημόσιες αρχές με τα αθλητικά κινήματα και κατά την άτυπη συνεδρία των Υπουργών του Ιουλίου μιλήσαμε πολύ για τις προσδοκίες του αθλητικού κινήματος με τον Επίτροπο Νοβράτητς και τους εκπροσώπους των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών. Πέμπτη πρωτοβουλία. Πρώτο προτεραιότητα. Θα ήθελα να σας πω ότι το Λουξεμβούργο τον Ιούλιο συνυπέγραψε μαζί με, τα άλλα 11, με άλλα 11 κράτη-μέλη μία διάσκεψη κατά της χειραγώγησης των ΣΥΚΕ αγώνων. Υπάρχει και η απόφαση του Συμβουλίου για αυτό το θέμα υπό τη Λετωνική Προεδρία και η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται. Η Προεδρία μας θα χειριστεί το θέμα αυτό με μεγάλη προτεραιότητα εφόσον συνυπογράφει και η Ένωση και τα κράτη-μέλη της μεμονωμένα αυτή την πρώτη διεθνή σύμβαση κατά των ΣΥΚΕ αγώνων. Θέλουμε αγώνες και αθλητισμό χωρίς ούτε ντόπινγκ ούτε πληρωμένους αγώνες. Τώρα οι οικονομικές επιπτώσεις του αθλητισμού αναγνωρίζονται από όλους. Το είπαν και οι προηγούμενες Ιταλική και Λετωνική Προεδρία. Τώρα που καταλήξουν αυτές οι συζητήσεις, τον Οκτώβριο στο Λουξεμβούργο η Προεδρία μας θα οργανώσει διάσκεψη με τίτλο η δημιουργία ανάπτυξης και πλούτου από τον αθλητισμό με εμπειρογνώμονες και του Συμβουλίου. Και για το παρόμοιο θέμα, για βιώσιμη ανάπτυξη του αθλητισμού, λαμβάνονται υπόψη και τα περιβαλλοντολογικά, οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία του αθλητισμού και θα συμμετάσχουμε ως Προεδρία στη διάσκεψη των Υπουργών που οργανώνουν Υπουργοί Αθλητισμού στη Γαλλία για την βιωσιμότητα, sustainability στα αγγλικά, των μεγάλων αθλη, διεθνών αθλητικών αγώνων. Διάσκεψη που διοργανώνεται στα πλαίσια της μεγάλης COP21 που οργανώνει η Γαλλία στο τέλος του έτους. Τέλος για να καταλήξω δύο μικρά σημεία. Η Προεδρία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη των πραγμάτων για την προστασία των δεδομένων και για τα τρόφιμα, την ενιαία ψηφιακή αγορά και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά την Κομισιόν αλλά και την Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή για τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού που θα συζητήσετε αν δεν απατώμε μετά. Σας ευχαριστώ πάντως για όσα θα πείτε και για τις ερωτήσεις που σίγουρα θα θέσετε. Και ελπίζω να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτές τις διασκέψεις που σας ανέφερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Ακούσαμε όλους αυτούς τους στόχους σας με τους οποίους και απολύτως συμφωνούμε. Θα συζητήσουμε την οικονομική αξία του αθλητισμού στη συνέχεια αλλά θα πρέπει τώρα οι συντάκτες εκθέσεων να λάβουν το λόγο να μας πούνε τι πιστεύω στον πρόγραμμα της ε, Προεδρίας. Οπότε θα δώσω τώρα στους συναδέλφους το λόγο πρώτα πρώτα στους ε, συντονιστάς που είναι εδώ για τρία λεπτά ο καθένας. Στη συνέχεια θα έχουμε έναν δεύτερο γύρο ερωτήσεων από τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Ε, πέντε λεπτά για σας ε, αφού τεθούν οι ερωτήσεις κύριε Υπουργέ. Ανάλογα με το πόσες θα είναι οι ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ σήμερα και μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητες σας στον τομέα του αθλητισμού. Ξεκινήσατε με τον ε, σχολικό αθλητισμό και τον αθλητισμό για, ακόμη και για πολύ μικρά παιδιά, στους παιδικούς σταθμούς κτλ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο τομέα αυτός, αν και αντιμετωπίζουμε ε, διαρκώς το πρόβλημα ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε έναν συντονιστικό κυρίως ρόλο. Ε, και θεωρώ ότι πρόκειται για έναν ε, ε, τομέα στον οποίο θα πρέπει να ενισχυθούν οι βέλτιστες πρακτικές. Στην πόλη μου, στο Ντίσσελντορφ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε αναπτύξει ένα μοντέλο σύμφωνα με το, με το οποίο κάθε μαθητής δημοτικού σχολείου από τη Δευτέρα Δημοτικού ε, ελέγχεται σε σχέση με τις ικανότητες στον αθλητισμό, ενημερώνονται για τις σχετικές συστάσεις και οι γονείς του και στη συνέχεια όλη αυτή η διαδικασία ξαναγίνεται στην 5η και 6η Δημοτικού. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική μέθοδος, ένα εξαιρετικό εργαλείο που μάλιστα έχει υιοθετηθεί ήδη από πάρα πολλούς δήμους και κοινότητες στη Γερμανία και νομίζω ότι μπορούμε να, παρατρύν, παροτρύνουμε και άλλα κράτη-μέλη να ε, υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο ακριβώς γιατί δεν είναι δυνατόν να μπορούν πάντοτε οι γονείς να έχουν πλήρη εικόνα για το ποιε είναι οι κανότες του παιδιού τους. Δεύτερο θέμα, ακαιρεότητα. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όχι μόνο σε σχέση με, την, με τον ντόπινγκ αλλά και σε σχέση με τα περιστατικά και τα συμβαίνοντα στην FIFA. Απαιτείται και εδώ η προώθηση της ακαιρεότητα, αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά το ντόπινγκ μήπως τελικά αποτελεί αυτό ο τομέας ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να αναλυφθούν νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ε, Γερμανία μάλιστα το ντόπινγκ έχει ενταχθεί και στον ποινικό ε, κώδικα, δεν αποτελεί πλέον μια απλή αστική ε, παράβαση αλλά ποινικό αδίκημα. Μήπως θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε να ρυθμίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα και σε ενωσιακό επίπεδο, μήπως θα έπρεπε να καταρτιστεί, να εκπονηθεί μια ευρωπαϊκή οδηγία. Τελευταίο θέμα, διπλές καριέρες. Διπλή καριέρα. Ε, πάντοτε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας εδώ στο Κοινοβούλιο, διότι ε, παρά τον ε, ενθουσιασμό που, που εμφανίζουν οι πρωταθλητές, ε, χρειάζεται πάντοτε να τους υπενθυμίζουμε και να επιθυμίζουμε και στους ανθρώπους ότι πρόκειται για μια καριέρα η οποία λύγει στα 35 το πολύ. Και χρειάζεται αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα και αργότερα δηλαδή να ζουν, να βιοπορίζονται, χρειάζονται εκπαίδευση γι' αυτό. Οπότε, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των ε, αθλητών και των πρωταθλητών, θα ήθελα να καλέσω ε, σε μια μη γραφειοκρατική μέθοδο χειρισμού του συγκεκριμένου ζητήματος που εμπεριέχει και την ε, αμοιβαία αναγνώριση των ε, εκπαιδευτικών ε, και των μορφωτικών των σπουδών του κάθε πρωταθλητή. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική βούληση προκειμένου να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Τα κράτη-μέλη δηλαδή θα πρέπει να φροντίσουν ώστε τα παιδιά να μην έχουν μόνο τη δυνατότητα να αθληθούν και να ε, παρακολουθήσουν κατάλληλη μόρφωση, αλλά θα πρέπει τα κράτη-μέλη από πριν να φροντίζουν και για την μετέπειτα σταδιοδρομία των αθλητών και των πρωταθλητών, γιατί δεν θα γίνουν όλοι προφανώς διαιτητές. Πρόκειται για μια ευθύνη που βαρύνει και τα κράτη-μέλη, αλλά και τους αθλητικούς συλλόγους και αυτή την ευθύνη δεν μπορούν να ε, την απαρνηθούν. Julie Ward Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε το θέμα του αθλητισμού. Η σημερινή συζήτηση. Ήθελα να σκεφτούμε λίγο ε, τη σύνδεση μεταξύ του ε, αθλητισμού και άλλων τομέων της ζωής. Ιδιαίτερα τη σύνδεση μεταξύ του αθλητισμού και του πολιτισμού, της τέχνης διότι ο χορός είναι μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης και ε, συνδέεται και με τον αθλητισμό. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί χορευτές που είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές για παράδειγμα. Και ο χορός πλέον ε, βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα αναλυτικά προγράμματα, στα σχολεία. Και ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν και ευρύτερε παράμετροι που αφορούν τον αθλητισμό και νομίζω ότι χρειάζεται να γκρεμίσουμε αυτά τα φράγματα. Στον αθλητισμό υπάρχει ανταγωνισμός και πολλές φορές ε, παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός ε, αυτό του δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αθλούνται και να έχουν φυσική δραστηριότητα. Υπάρχει και ένα ευρύτερο θέμα που σχετίζεται με το πώς ε, λειτουργούν ε, οι σύλλογοι και οι αθλητικές ομάδες και το πώς έχουν αντιμετωπίσει το bullying. Όπως για παράδειγμα μέσω του Rainbow Laces που ε, ασχολείται με την καταπολέμηση της ομοφοβίας. Είναι μια εκπληκτική εκστρατεία που διοργανώθηκε στην χώρα μου. Και είμαι και πολύ περήφανη που έχουμε και την πρωτοβουλία «Δείξτε κόκκινη κάρτα στο ρατσισμό» που ξεκίνησε από τον ποδοσφαιρικό όμιλο του Σάντερλαντ που και πλέον έχει αποκτήσει πανεθνικά χαρακτηριστικά η εκστρατεία αυτή και νομίζω ότι θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για σας να τονίσετε τους τομείς στους οποίους ο αθλητισμός δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να σκεφτούν ευρύτερα. Τι σημαίνει για για τους, ε, για τους ανθρώπους. Τι σημαίνει η συμπερίληψη, η, ε, η, ε, η, καταπολέμηση των αποκλεισμών. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ και στους γερμανικούς ποδοσφαι... στις ομάδες ποδοσφαίρου από τη Γερμανία και τις, ε, τα πανό που αναρτήθηκαν στα γήπεδα που ε, καλωσόριζαν τους πρόσφυγες. Θέλω να πω ότι ο αθλητισμός πολλές φορές μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα που οι πολιτικοί δεν μπορούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε με ναι, μεγάλη μας ευχαρίστηση ακούσαμε τα όσα έχει να μας πει ο Υπουργός. Πρώτα πρώτα να σας πω ότι συμφωνώ με όσα πρότεινα. Και για το πώς θα εκπαιδεύσουμε άντρες και γυναίκες στον αθλητισμό. Είναι πολύ σημαντικό ε, αυτή η δυτή σταδιοδρομία, δηλαδή θεωρητική κατάρτιση και πρακτική ασχόληση με τον Και επίσης να υπάρχει δυνατότητα κινητικότητας. Συμφωνώ με την ε, συνάδελφο Πέτρα, αν υπάρχει αυτή η κινητικότητα, τότε υπάρχει αυτόματα η αμοιβαία αναγνώριση και της ε, θεωρητικής γνώσης. Βέβαια πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι και κινητικότητα δεν μπορεί να είναι μόνο κινητικότητα για τους αθλητές αλλά και για τους προπονητές. Και αυτοί θα πρέπει να μπορούν να μετακινηθούν και να κινηθούν. Κάτι άλλο τώρα. Ο σημαντικός ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση των ανηλίκων. Από προσωπική μου εμπειρία γνωρίζω ότι το καλύτερο που μπορεί κανείς να έχει λύσει προβλήματα των παιδιών ακόμα για τη βία μεταξύ των παιδιών είναι αθλητισμός. Κάποιος δηλαδή πάρα πολύ γνωστός ας πούμε αθλητής του τζούντο θα διδάξει στα παιδιά στο πώς θα κατευθύνουν την ενέργειά τους αλλού και όχι στο να βλάπτουν κάποιον άλλο. Νομίζω αυτή είναι πάρα πολύ καλή ιδέα και ίσω θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα και έτσι να μπορέσουμε και να καλέσουμε και από του γνωστού αθλητέ και αθλήτριε. Ο αθλητισμό είναι κάτι το καθαρό, κάτι το καλό. Αυτό μπορεί να καταπολεμήσει και τη χρήση ναρκωτικών. Άρα κανεί μπορεί να πετύχει πολλά να μετά. τα μετά. Λουίτζι Μόργαν. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Πραγματικά θεωρώ ότι αυτές οι πέντε προτεραιότητες που τάξατε είναι σημαντικό στοιχείο ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη πολιτική για τον ε, αθλητισμό. Εγώ έλαβα το λόγο γιατί νομίζω ότι η προσοχή που δίνουμε είναι ο αθλητισμός σε επίπεδο ανταγωνισμού. Όμως χρειάζεται να γίνει ε, ευαισθητοποίηση και των ανηλίκων στον αθλητισμό και σε αυτή την τρυφερή ηλικία και έτσι να μπορέσουμε καλύτερα να ε, διαδώσουμε αθλητισμό. Ε, να έτσι να τους ελκύσουμε την προσοχή και να έχουμε επομένως ε, μία προώθηση του αθλητισμού που δεν είναι ανταγωνιστικός. Όλοι νομίζω συμφωνούμε πάνω σε αυτό και δεν θέλουμε επομένω να πάρουν άλλη κατεύθυνση προσπαθίες μας. Έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν βρίσκω εδώ το όνομά σας. Α, είναι ο κύριος Βούκοβιτς, ο επικεφαλής σχετικής υπηρεσίας. Α, όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, γιατί ένας άλλος, άλλος ο κύριος Τάκουλα έχει δει το λόγο. Κατόπιν, Επιτροπή. Τάκουλα. Χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι εδώ επί από δέκα μήνες και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι εκ μέρους της Άλντε. Γνωρίζουμε ότι ο αθλητισμός είναι εξαιρετικό εργαλείο στην ε, καταπολέμηση της παχυσαρκίας, της, του διαβήτη τύπου 2 και άλλων ασθενειών και προβλημάτων υγείας. Το πρόβλημα είναι όμως ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι αρμοδιότητες μας είναι περιορισμένες. Τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που έχουν την αρμοδιότητα στον τομέα του αθλητισμού. Φυσικά μπορούμε να ενθαρρύνουμε και να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν τα σωστά. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον Υπουργό ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβετε στη διάρκεια της Προεδρίας σας σε συνεργασία με... και στις συναντήσεις που θα έχετε με τους συναδέλφους σας υπουργούς από τα άλλα κράτη-μέλη. Υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι. Α, έχει εσείς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να τοποθετηθώ για τις παρατηρήσεις σε γενικό επίπεδο από πλευράς Επιτροπής. Θεωρούμε πάρα πολύ θετικά όλα αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος ε, Υπουργός και όσοι έλαβαν ε, τον λόγο για την ε, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα του Αθλητισμού. Δεν θέλω να επεκταθώ και να πολυλογήσω, αλλά τα πρώτα να δείχνουν στο ότι ήταν πολύ πετυχημένη η πρώτη στόχη και ότι αυτή η εβδομάδα πρόκειται μακροπρόθεσμα να συμβάλλει όσον αφορά την προώθηση της αθλητικής δραστηριότητας στα κράτη-μέλη. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο, κάτι για την Λουξεμβουργική Προεδρία, γιατί νομίζω ότι όλα τα σημεία κλειδιά θίξατε κύριε Υπουργέ, όλα αυτά που μας έχουν απασχολήσει και θα συνεργαστούμε μαζί σας και με το Κοινοβούλιο. Όμως, ε, να σας ε, αναφέρω και εγώ κάτι για τους ΣΥΚΕ αγώνες. Ο Επίτροπος Ναύρατσετς έχει δεσμευτεί να ασχοληθεί, να καταβάλει προσπάθειες προς εκείνη την κατεύθυνση και να συνεργαστεί πάνω σε αυτό με τα κράτη μέλη, αλλά και για τον τοπάρισμα. Είμαστε στο πλάι της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας. Για να δούμε τι γίνεται σε σχέση με το ψήφισμα του 2011 ε, και επίση η διπλή σταδιοδρομία είναι θέμα επικαιρότητα. μια που τώρα είμαστε σε συγκυρία κρίσεω. είχε επισημανθεί η διπλή σταδιοδρομία σαν κάτι βασικό που θα πρέπει να απασχολήσει την Επιτροπή κάνουμε τώρα μια μελέτη και θα την υποβάλουμε προσεχώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με κάποιες σκέψεις μας για προβληματισμό. Επίσης όσον αφορά την διακυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι δεν μπορέσαμε εδώ να τα καλύψουμε όλα. Βεβαίω θα πρέπει να δούμε ε, μετά τόσο έγινε στους τελευταίους μήνες ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 14-17 που ενέκρινε το Συμβούλιο αλλά έχουμε και εμείς έναν ρόλο. Η διακυβέρνηση επομένως σε αυτό το πρόγραμμα είναι μία από τις πέντε προτεραιότητες. Καλύπτονται διάφορες ιδέες των ε, εμπειρογνωμόνων οπότε ε, σε επόμενες εβδομάδες πρόκειται να ε, επανέλθει σε αυτό ο Επίτροπος σε επαφή με το Κοινοβούλιο. Δεν τα θίξαμε όλα, αλλά ό,τι θέλετε να το προσθέσουν. Ευχαριστούμε λέει πρόεδρο. Αν περιμένουμε κάποιον άλλο συναδελφό σας. Αλλά πάντως είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Στα πλαίσια των ομάδων εργασία. Και τώρα είναι σημαντικό να σε αυτούς τους συναδέλφους κύριε Υπουργέ γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει ε, αποκλειστική κοινωτική αρμοδιότητα όπως είπε ο συνάδελφος όμως ε, έχουμε κάποιες κοινέ διατάξεις κάτι το, το, το ζητήσαμε και είπαμε θα πρέπει να γίνει νομοθετική προσπάθεια και Γι' αυτό και θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρωτοβουλία, την οδηγία για τον τοπάρισμα και επίσης το άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των, των ΣΥΚΕ αγώνων αλλά και η διπλή σταδιοδρομία ήταν σημαντικό που αναφέρθηκε όσον αφορά την αντιστοιχία αθλητισμού και σταδιοδρομίας. Είμαι βέβαιο ότι με αυτές τις προτεραιότητες μας αναφέρατε πρόκειται να υπάρξει πρόοδος στο Συμβούλιο και με την ευκαιρία όμως της διάσκεψης που αναφέραμε. Έχετε το λόγο. Euh, euh, Ο Υπουργό, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όσοι έλαβαν το λόγο. Μπορώ να συνοψίσω λέγοντά σα ότι εδώ νιώθω σαν στο σπίτι μου γιατί πολλές φορές μιλώντας για τον αθλητισμό είτε σε διεθνές ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό θεωρείται κάτι, κάτι περίεργο, σαν να μην ήταν στοιχείο πολιτιστικό. Όχι, έτσι καλά το πήγαμε εδώ, είναι ωραίο εδώ. Και γι' αυτό και σας ανέπτυξα έτσι ότι αθλητισμός δεν είναι μόνο μάτς και ανταγωνισμός. Υπάρχει προσθεμένη αξία, πολλές φορές δεν μπορούμε καν να την υπολογίσουμε. Είναι το ευζήν, είναι η κοινωνική ένταξη, είναι κάποιες αξίες που προκύπτουν. Και αντιστοιχεί με τις άλλες πολιτικές, πολιτικού του αθλητισμού. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε διάφορα προγράμματα. Αλλά εδώ στη δική σας επιτροπή ε, είναι σωστό, θέλετε να προωθήσετε τον αθλητισμό και να αναδείξετε τις σχετικές αξίες πέραν του ανταγωνισμού. Αυτό για να ξεκινήσω, για να θέσω έτσι ένα πλαίσιο τρόπο όσον αφορά τις επιμέρους ερωτήσεις αλλά και τις επιμέρους θετικές σκέψεις. Πρώτα απ' την κυρία Κάμερβερτ στα γερμανικά και να συνεχίσω στα γερμανικά. Γνωρίζετε ότι το σημαντικό είναι αυτά τα πρακτικά παραδείγματα. Αυτό θέλουμε και εμείς ως Προεδρία. Τις βέλτιστες αυτές πρακτικές. Ίσως να μπορέσουμε να καταρτήσουμε και έναν κατάλογο για να μπορούμε να βλέπουμε ποια εγχειρήματα, ποιες προσπάθειες με παιδιά έχουν γίνει, ποιες έχουν στεφτεί με επιτυχία. Παιδιά ακόμη και κάτω των 5 ετών, αυτό χρειαζόμαστε. Συνεργασίες, συνέργειες. Να μην λέμε δηλαδή ότι όλα αυτά γίνονται απλά μόνο στις ομάδες και στους ε, συλλόγους και στα σχολεία. Χρειαζόμαστε και άλλους φορείς που θα συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία τους παιδικούς σταθμούς, τους γονείς, εκεί που ζουν τα παιδιά. Εκεί χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα προωθήσουν τον, τον αθλητισμό και θα προσφέρουν στα παιδιά την, ε, να ζήσουν μια ζωή που συστατικό στοιχείο της θα είναι ο αθλητισμός. Και εδώ, ε, σε ό,τι αφορά το, την ακαιρεότητα, το στήσιμο των παιχνιδιών και το ντόπινγκ είναι πάντοτε ζητήματα που σχετίζονται με την κακή διακυβέρνηση δεν φαίνονται πάντα αυτά τα φαινόμενα, αλλά στο ντόπινγκ πρέπει να κάνουμε περισσότερο. Δεν αφορά, αυτό πρέπει να πούμε και στους νέους ανθρώπους, δεν αφορά μόνο το ντόπινγκ το ζήτημα της ακαιρεότητας, αλλά και την υγεία σας. Είναι ένα θέμα όπου ο αγώνας δεν θα τελειώσει ποτέ, διότι κάθε φορά υπάρχουν νέα μέσα, βλέπετε, που προσπαθούν διάφοροι επιτίδοι ακόμα και με μικρές, πολύ μικρές δόσεις να συνεχίσουν αυτή την κατάσταση με τη φαρμακοδιέγερση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και σε αυτό το τομέα ευρωπαϊκή συνεργασία. Και στο ερώτημά σας αν ίσως θα πρέπει να αναλευθούν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, η απάντηση είναι σαφώς ναι. Και διεθνώς. Και θα πρέπει το κεκτημένο που υπάρχει να εφαρμοστεί σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και από εκεί και πέρα να εξετάσουμε ποια περιθώρια και ποιες δυνατότητες υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να το εξετάσουμε για να το... Αν, αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα δηλαδή και πώς θα το κάνουμε. Στο τελευταίο ζήτημα που θέσατε θα ε, όσον αφορά την μετέπειτα σταδιοδρομία των αθλητών ε, θα, θα μιλήσω αργότερα. Και τώρα να συνεχίσουμε αυτά που είπε η κυρία Βόρτ που μας ε, είπε για τον αθλητισμό πέραν του ανταγωνισμού. Όχι, για μένα δεν είναι σπουδαίο, δεν είναι σημαντικό να κάνει κανείς ανταγωνιστικό σπορ. Θα μπορεί κανείς να κάνει χορό, γιατί υπάρχουν ε, ε, το τι κάνει ο καθένας ατομικά ούτως ώστε να προάγεται η κίνηση και ο αθλητισμός, η αθλητική κίνηση. Βεβαίω και θα πάνω απ' όλα ε, είναι το να κινείται κανεί με οποιοδήποτε τρόπο, ε, κυρία Αγόρ. Και ε, ακριβώ η σχετική θεματική είναι πολύ σημαντική. Και έτσι έχουμε και την κοινωνική ολοκλήρωση και την κοινωνική ένταξη σε όλες τις χώρες. Είναι η ιδιώδης πλατφόρμα αθλητισμός για να συμμετέχει κανείς και καν για ένταξη, μιλάω για συμμετοχή. Για να μπορεί κανείς να εμπλακεί στο κοινικό γίγνεσθε μέσω αυτής της συμμετοχής. Τώρα ε, είχαμε την ερώτηση κυρίας Λιμπάτσκα που είπε κάτι πολύ σημαντικό. Μίλησε για την διπλή σταδιοδρομία σε σχέση και με την κινητικότητα. Έτσι η Ευρώπη έγινε πιο μεγάλη με αυτή την ελευθερία κίνησης. Αυτό είναι σημαντικό και από αθλητικής πλευράς και εκπαιδευτικής. Πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα να καταλήξουμε σε κάποια κοινά προγράμματα. Προγράμματα εκπαιδευτικά που να μην αφορούν μόνο την διπλή σταδιοδρομία αλλά να αξιοποιούν τον αθλητισμό και τους αθλητές κατά την επαγγελματική σταδιοδρομία και μετά. Γιατί ακριβώς αυτοί οι επαγγελματίες αθλητές έχουν μια μικρή διαδρομή και μετά όμως θα πρέπει κάτι να γίνεται για να συνεχίζουν τη ζωή τους. Τώρα, γι' αυτό που μας είπε ο κύριος Μοργάνο και αυτός ανέφερε πόσο σημαντικές είναι διάφορες διαργανώσεις και όχι μόνο οι ανταγωνιστικές αλλά και την αθλητική πτυχή, ποδόσφαιρο, ποδηλασία αλλά και πέραν αυτών έχουμε και άλλα σπορ πάρα πολύ σημαντικά και είδα γίνεται το σημαντικό βιβλίο στην αρχή της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για το τι γίνεται σε κάθε χώρα Πόσο εύκολα μπορεί κανείς να κάνει διάφορα σπορ χωρίς να ξοδεύει πολλά χρήματα. Απλώς ε, κανείς ε, μπορεί ε, έτσι να παίζει, να δημιουργεί αθλητικά. Ναι, ναι, συμφωνώ και είμαι στο δικό σας μήκος κύματος. Κύριε Τάκουλα, για να ολοκληρώσουμε για το πώς θα γίνει η ενημέρωση των συναδελφών. Νομίζω ότι υπάρχει το σχετικό εργαλείο. Πολύ σημαντικό. Αυτή η πρώτη εβδομάδα αθλητισμού στην Ευρώπη. Θα κάνουμε έναν απολογισμό, μια έκθεση, αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να έχουμε αυτή την εβδομάδα κινητικότητα. Τώρα αυτό έχει θεσμικό χαρακτήρα παντού, σε όλε τι χώρε. Να αξιοποιήσουμε επομένω αυτή την πρωτοβουλία για να δείξουμε την ποικιλία του αθλητισμού και τη συνέπεια των επιμέρους πολιτικών που θα πρέπει να συνάδουν μεταξύ τους των ε, εθνικών πρακτικών και δεν για το Λουξεμβούργο, το λέω απλώς σε παρένθεση, έχουμε εκεί πέρα ε, με ένα πρόγραμμα που λέγεται ε, τρώτε γινότερα, κινηθείτε περισσότερο και όλα τα υπουργεία του Λουξεμβούργου έχουν εμπλακεί σε αυτό το πρόγραμμα. Να, τι εννοούμε συνεκτικές πολιτικές και ενημέρωση του κόσμου. Καλή πρακτική. Να ποια τα μέσα και τα εργαλεία για να τα καταφέρουμε. Και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η πρόεδρος για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Να συνεχίσουμε τον διάλογο με το Συμβούλιο, με την Προεδρία, εμείς ως Επιτροπή, γιατί αυτές σας οι προτεραιότητες θα πρέπει να μας απασχολήσουν καθήκον μας. Και θα έχουμε και αυτήν την διάσκεψη που είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Τώρα κάτι άλλο, εγώ σαν Ιταλίδα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, αυτή η εικόνα. Έχουμε αυτές τις δύο Ιταλές νέες, την Πενέτα Βίντζε που απαιτέλσαν ένα παράδειγμα προς μίμηση στο US Open, στο τέννις. Τον είπα γιατί ακριβώ λέμε και για κάποια ε, σπορ, που και τις γυναίκες. Ήταν επομένως αυτή η εικόνα πάρα πολύ όμορφη. Ήταν ε, μια ε, εικόνα υγιούς ανταγωνισμού, φιλίας, τρυφερή εικόνα. Επομένως δεν έχουμε μόνο την παθολογία του αθλητισμού, έχουμε και την εκπαιδευτική πλευρά. Σας ευχαριστούμε και καλή επιτυχία για την Προεδρία σας. I think it's a workshop now. Yeah, okay, so I. Uh, Παρακαλώ να έρθουν οι εμπειρογνώμονες για να αρχίσουμε τη συνέχεια. Bene, allora, και τώρα αρχίσουμε με το δεύτερο τμήμα της τη διάταξη. Είναι ήδη εδώ οι εμπειρογνώμονε. Παρακαλώ, ελάτε. Welcome ορίσατε όλοι. Ευχαριστούμε τους εμπειρογνώμονε μας που ήρθαν εδώ. Σας ευχαριστούμε. Μας τιμά η παρουσία σας. Όπως γνωρίζετε, το έχετε, έχετε αυτό το σημείο, το έχετε ακουστικά. Σήμερα θέλουμε να προβληματιστούμε πάνω στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Έχουμε αυτό το εργαστήριο από το τμήμα πολιτικής του Κοινοβουλίου. Ετήσι της Επιτροπής μας. Μιλούμε για 1.020 αθλητές, μιλούμε για 30 χώρες που έχουν συμμετάσχει και όλοι αυτοί είναι πρεσβευτές του αθλητισμού. Πρόκειται για κάποιους αθλητές. Και επομένως έχουμε μια μεγάλη πρωτοβουλία για να στηριχτεί αυτή η εβδομάδα του αθλητισμού και να πράγμα τον αθλητισμό και την αθλητική δραστηριότητα, διαφορετικό τρόπο ζωή, πολύ σημαντικό για την ε, κοινωνική ένταξη. Είχαμε και τον Υπουργό πράγμα που μα έλεγε τι γίνεται ε, όσον αφορά την συμμετοχικότητα που θεωρούμε ότι αυτό θα είναι ο καρπός αυτής της πρωτοβουλίας. Οπότε Είδαμε τις, ε, ότι σωστά του κοινό πανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία και σε σχολεία, σε πόλεις, σε διάφορους φορείς ε, είχαμε διάφορες εκδηλώσεις με πολλά θέματα και ε, ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε μια αξιολόγηση αυτής της εβδομάδας πρώτα πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπροσωπήθηκε η Επιτροπή από τον επικεφαλής της σχετικής υπηρεσίας. Και θα ήθελα επίσης να σας πω σε σχέση με την ακρόαση του Υπουργού του Λουξεμβούργου ότι επιβιώνεται πως αυτά τα θέματα τα οποία για σήμερα διαλέξαμε είναι θέματα τα οποία αποτελούν προτεραιότητες της ε, Λουξεμβουργιανής Προεδρίας αλλά ε, αναφέρονται και στο πρόγραμμα εργασιών του Συμβουλίου. Άρα έτσι προχωρούμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Ε, τα αναφέρουμε ποια είναι πρώτα πρώτα την ακεραιότητα στον αθλητισμό. Ευχαριστούμε αυτούς που ήρθαν γιατί έχουν συμμετάσχει σε αυτήν την ε, εβδομάδα. Επίσης έχουμε τον David Walsh, ε, περίφημο δημοσιογράφο των Sunday Times που θα μας μιλήσει αυτό το ζήτημα της ε, ακαιρεότητας. Και επίσης θα μας μιλήσει για την καλή διακυβέρνηση. Θα μας πει για τις έρευνες που έχει κάνει όσον αφορά τον Τοπάζ στην ε, ποδηλασία σε σχέση με τον Άμστρον και την Postal Service, μια ομάδα αμερικανική. Κατόπιν θα έχουμε έρωτα απαντήσει προς και από τον κύριο Γουόλς για ένα δεκάλεπτο και μετά θα συνεχίσουμε με τις άλλες ε, εισηγήσεις όσον αφορά πρώτα πρώτα ε, τον αθλητισμό, σε σχέση με τη δημιουργία ανοιχτή και κοινωνίας που δεν αποκλεί κανέναν από τον καθηγητή Χένρι ο οποίος ε, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Λάφπορο. Επίσης μετά έχουμε την οικονομική διάσταση του αθλητισμού που απεσχόλησε και την πλούσια ε, Βαργίνη Προεδρία. Θα μας μιλήσει η, η δόκτωρ Άννα Κλάσνερ που είναι αναπληρωτής διευθύντρια του Sportsecon Austria ενός ε, αθλητικού ιδρύματος. Και θα έχουμε 15 λεπτά ερωταπαντήσεις, οπότε και τότε θα λάβει τον ε, λόγο ο επικεφαλής ε, της ε, αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής, ο κύριος Ιβ Λέλοστεκ. Νομίζω ότι όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ ε, ενδιαφέροντα και κατόπιν θα έχουμε ένα γυρό τραπέζι από τους φορείς που έχουμε προσκαλέσει. Οπότε ευθύ αμέσω, κύριε Βόλς, σας δίνω τη σκητάλη. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που μου επιθύνατε αυτή την πρόσκληση να έρθω και να σας μιλήσω. Την αποδέχτηκα με μεγάλη χαρά γιατί είμαι αθλητικογράφος εδώ και 37 χρόνια και έχω περάσει τα τελευταία 15-16 από τα 22 χρόνια, τα προηγούμενα δηλαδή, θέλοντας να γίνω αθλητικογράφος. Ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα να γίνω στη ζωή μου και νομίζω ότι δεν θα σταματήσω ποτέ όσο ζω να είμαι αθλητικογράφος. Αλλά όχι με τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησα να εργάζομαι, να ασχολούμαι με την αθλητικογραφία. Ήμουν παιδί, ήμουν 10 χρονών, ζούσα σε μια μικρή πόλη στην Ιρλανδία και ξυπνούσα σε 7 το πρωί και το μόνο που θυμάμαι είναι να θέλω να διαβάσω την ε, εφημερίδα. Δεν μπορούσα να περιμένω μέχρι να ανοίξει το μαγαζάκι της Jack, ε, το μαγαζάκι της γειτονιάς μου και το γαλατά που έφερνε μαζί με το γάλα τις ε, εφημερίδες που τις άφηνε έξω από το μαγαζί και εγώ περίμενα, προσπαθούσα από τον πάκο των εφημερίδων να βγάλω μία για να διαβάσω τις αθλητικές σελίδες. Αυτό ήταν, αυτό ήθελα να γίνω στη ζωή μου. Ξεκίνησα στο επάγγελμα ως ένας φίλαθλος με γραφομηχανή. Ήμουν φίλαθλος που κατάφερε να βγάλω τα, τα χρήματά μου από το πάθος μου. Η οπτική μου άλλαξε με τα χρόνια. Μπορεί να αναρωτιέστε γιατί. Η απάντηση είναι απλή. Πήγα στη Σεούλ το 1988. Ήταν η πρώτη μου Ολυμπιακή αγώνας. Μπεν Τζόνσον εναντίον Καρλ Λιούις θα είχαν την ε, σημαντικότερη, τον σημαντικότερο αγώνα στην ιστορία ε, του αθλήματος. Ήθελα να κερδίσει ο Μπεν Τζόνσον γιατί ήταν ε, outsider και θα, ενώ ο Καρλ Λιούις ήταν ο μεγάλος Αμερικανός, ο Μπεν Τζόνσον ήταν Καναδός. Εγώ, ο, ο με την ε, γραφομηχανή, ήθελα τον Μπεν Τζόνσον και στις 3 το πρωί, δύο μέρες μετά, κάποιος χτύπησε την πόρτα μου. Συνήθως αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Άνοιξα την πόρτα και μου είπαν ότι ο Τζόνσον αποδειχθήκε ότι είχε το παριστεί. Αυτό άλλαξε τη στάση μου. Παρότι στεναχωρέθηκα, προσπάθησα να το εξαρθολογήσω, να πω ότι εντάξει ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση και τα λοιπά. Πήγα στο Sunday Times το 1996. Είχα δουλέψει ως αθλητικογράφος σε Ιρλανδικές εφημερίδες μέχρι τότε. Ε, κάλυψα έναν αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης. Πήγα στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα. Και ένας από τους πιο διάσημους ε, αθλητές ήταν ένας 26χρονος ε, κολυμβητής, Ιρλανδός. Είχαμε κερδίσει μέχρι τότε ως χώρα μόνο τέσσερα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαμε και ένα αστείο που λέγαμε στην Ιρλανδία, ότι αν ο κολυμβητής μας δεν πνιγόταν τότε θα ήταν καλό. Και εκείνη την, ε, σε εκείνη τη φάση είχαμε τρία χρυσά μετάλλια μέσα σε μια εβδομάδα. Υπήρχαν σοβαροί λόγοι για να αμφιβάλλει κανείς για την ακαιρεότητα της όλης υπόθεσης. Και όταν εξέτασα εγώ από κοντά την υπόθεση δεν πίστεψα αυτά που έβλεπα. Με τρεις άλλους συναδέλφους είπαμε ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν ε, μπορούσε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πράγματι, η κολυμβήτρια εκείνη τελικά της αφαιρέθηκαν τα μετέλεια. Και να σας πω και μια προσωπική ιστορία που με επηρέασε σημαντικά στη ζωή μου και θα ήθελα να την ακούσετε σοβαρά όσον αφορά τη σχέση σας με τον αθλητισμό. Είναι μια ιστορία που σχετίζεται με τον θάνατο ε, του 12χρονου γιού μου. Από αυτοκίνητο ε, οδηγούσε το ποδήλατο και τον χτύπησε αυτοκίνητο. Αποφασίσαμε ως οικογένεια να το συζητήσουμε να μιλούμε για τον Τζον, τον γιο μου και να υπενθυμίζουμε και στους γύρω μας τι σήμαινε για μας αυτός. Και ε, ως πατέρας του Τζον, αυτό που ήθελα να κάνω είναι να μάθω πράγματα για εκείνον που δεν τα γνώριζα. Πήγα στον, στον προπονητή του, του ποδοσφαίρου, του ράγμπι, πήγα, μίλησα με τους δασκάλους του. Και ένα από του δασκάλου του μου είπε μια εξαιρετική ιστορία. Μου είπε ότι όταν ο Τζον ήταν 7 ή 8 χρονών, και διάβαζαν ε, την ιστορία του μικρού Ιησού για την ε, Ιωσήφ και την Μαρία που ε, κατάφεραν να βρουν επιτέλους μια φάτνη, ένα στάβλο στον οποίο γεννήθηκε το παιδί τους ο Ιησούς και ήρθαν τρεις ε, μάγοι που τους δίνουν τα δώρα και η Μαρία και ο Ιωσήφ επιστρέφουν εκεί από που προέρχονταν και ζήσαν μια λιτή και ταπεινή ζωή γιατί ο Ιωσήφ ήταν ένας ταπεινός ξυλοκόπος και τότε ο Τζον ε, σήκωσε το χέρι του και είπε «Κυρία, είπατε ότι η Μαρία και ο Ιωσήφ δεν είχαν πολλά και τι έκαναν τελικά με εκείνο το χρυσό που, του είχαν, που τους είχαν φέρει οι τρεις μάγοι» και του είπε «Τζον, διαβάζω αυτή την ιστορία εδώ και 33 χρόνια και ποτέ κανένα παιδάκι δεν με έχει, ε, ε, με έχει ρωτήσει αυτό το πράγμα και ειλικρινά δεν ξέρω. Όταν η δασκάλα του μου είπα αυτό το πράγμα, συνειδητοποίησα ότι ακριβώς αυτό είναι το κέντρο, ο πυρήνας της δημοσιογραφίας, ακόμη και αν το βασικό, το, το προφανές. Ακόμη και αν σε κοροϊδέψουν. Και αποφάσισα ότι έτσι θα συνέχιζα. Θα έθετα τα προφανή ερωτήματα. Είμαι γνωστός στους δημοσιογραφικούς κύκλους ως εκείνος που δεν πίστευσε ποτέ τον Λάρντς Άρμστρομ που προσπάθησε να πει στον κόσμο ποια είναι η αλήθεια. Και με ενέπνευσε η ερώτηση που έκανε ο γιος μου όταν άρχισα να ασχολούμαι με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και από τη δική σας σκοπιά το ερώτημα που πρέπει να θέτετε είναι αν ο Λάντς Άνστρονγκ έπαιρνε ντόπινγκ από την αρχή πώς έγινε και χρειαστήκαμε 13 χρόνια μέχρι να μάθουμε την αλήθεια. Γιατί σας το λέω, το 1999 τη δεύτερη εβδομάδα της πρώτης Tour de France του Λάντς Άνστρονγκ ήταν σαφές ότι ο άνθρωπος παραβίαζε τους κανόνες. Δεν χρειαζόταν, δεν χρειαζόταν ε, να κάνει κανείς μεγάλη έρευνα δημοσιογραφική. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν κοινή λογική. Εδώ βλέπεις έναν καινούριον ε, ε, αθλητή που δεν έχει ποτέ συμμετάσχει. Φαινόταν καθαρός, η έλεγε ότι ήταν καθαρός. Όλοι γνώριζαν, η ελ άκουγαν τον ίδιο να λέει ότι δεν παίρνει φάρμακα και Υπήρχε ένας νέος αθλητής λοιπόν, ο κύριος Καθαρός. Ποιος ε, όμως τον τραμπούκιζε, ο Λαντς Άρμστρον. Υπήρχαν πάρα πολλοί λόγοι για να πιστέψει κανείς και να δει ότι πράγματι ο άνθρωπος αυτός έλεγε ψέματα. Γιατί μας πήρε όμως 13 χρόνια. Γιατί οι άνθρωποι που ήταν αρμόδιοι και δεν εννοώ μόνο ε, τους ε, φορείς διακυβέρνησης της εννοώ και τις τηλεοράσεις, τους δημοσιογράφους, τους χορηγούς, Φυσικά, είναι προφανέ ότι δεν θέλουν να χρηματοδοτούν αθλητέ που είναι διεφθαρμένοι, αλλά όλοι κάναν τα στραβά μάτια. Είχαν όλοι διαφορετικού λόγου και οι περισσότεροι από αυτού του λόγου σχετίζονταν με οικονομικά συμφέροντα. Για τι εφημερίδε, ήταν ωραία ε, υπόθεση, οι χορηγοί βγάζαν λεφτά, οι τηλεοράσει το ίδιο και ε, η διεθνή Ομοσπονδία Ποδηλασίας είχε έναν εξαιρετικό αθλητή που μπορούσε να τον πουλήσει. Γι' αυτό και δεν γίνονταν οι απαραίτητοι έλεγχοι για τον συγκεκριμένο αθλητή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε τη σημασία αυτού που έγινε με τον Lance Armstrong. Από το 1999 έως το 2005 δεν υπάρχει νικητής της Tour de France. Την τελευταία φορά που αυτό δεν είχε γίνει, για 7 χρόνια δηλαδή να μην έχουμε νικητή στην Tour de France, ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Αυτό έκανε το ντόπινγκ στο Tour de France. Αφαίρεσε τον ίδιο αριθμό ετών με νικητές όσο και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Μπορεί κανείς να πει ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Μπορεί να, είναι, να, να, να το σκεφτεί κανείς ως θηρίο πόσες φορές και να του κόψουμε το κεφάλι, αυτό ξαναβγαίνει. Και μπορεί να θεωρείται ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε. Κατά τη γνώμη μου, εσείς είστε οι πιο σημαντικοί άνθρωποι. Εσείς είστε αυτοί που μπορείτε να ξεκινήσετε τις πραγματικές αλλαγές που χρειαζόμαστε. Και ένας άλλος λόγος για τον οποίο αμφέβαλα για τον Λάντς Άρμστρομ ήταν το γεγονός ότι πριν από ένα χρόνο, ένα χρόνο νωρίτερα, ένα χρόνο πριν, οι τελωνιακές αρχές στη Γαλλία είχαν πει ότι θα κάνουν έρευνες στο ε. συγκεκριμένο ζήτημα διότι δεν υπάρχει μηχανισμός αυτορύθμισης στον τομέα της ποδηλασίας και θα τους βοηθήσουμε εμείς ώστε να απαλλαγούν από κάθε απάτη. Φυσικά δεν μιλάω και δεν θέλω να μιλήσω μόνο για την ε, ποδηλασία. Έχουμε και τη FIFA που εδώ και χρόνια όλοι γνωρίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αν το πάμε και λίγο παραπέρα, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει διαφθορά. Και παρόλα αυτά φαίνεται ότι είναι υπεράνω του νόμου. Αλλά δεν είναι. Υπάρχει μια έρευνα από την Ελβετία, από τις ΗΠΑ και ξαφνικά η FIFA κάνει λόγο για σοβαρές αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν. Μπορεί κανείς να πει μεταφορικά ότι αυτό έγινε με το πιστόλι στον κρόταφο. Αυτό ακριβώς έγινε πράγματι αλλά χρειάζεται οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι να λαμβάνουν τέτοιου είδους αποφάσεις. Συμφωνώ απόλυτα με την κίνηση να καταστεί σε όλες τις χώρες το ντόπινγκ ποινικό αδίκημα, διότι ο βαθμός εξαπάτησης, απάτης, ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ε, ευρώ. Σε κανέναν άλλο τομέα της ζωής δεν θα επιτρέπαμε σε ανθρώπους να κλέβουν τόσα πολλά χρήματα. Και να πω και κάτι που κολακεύει τις ε, κυβερνήσεις και τους πολιτικούς. Είμαι αθλητικογράφος, καλύπτω εκδηλώσεις αθλητικές και το, την υπόθεση του anti-doping. Ξέρετε ε, ότι πώς, πώς ορίζεται ο πρόεδρος της υπηρεσίας anti-doping. Πρώτα, ε, το, τη μία φορά τον ορίζουν οι κυβερνήσεις και την επόμενη φορά την τον ορίζει η Διεθνής ε, Ολυμπιακή Επιτροπή. Εγώ Χαίρομαι κάθε φορά που έχουμε πρόεδρο που έχει οριστεί από τις κυβερνήσεις γιατί ε, είναι πολύ πιο πιθανό αυτός να καταπολεμήσει τον ντόπινγκ και να μην υποχωρήσει σε πολιτικές πιέσεις. Κάτι που είναι παράδοξο, γιατί το αντίθετο θα περίμενε κανείς. Υπάρχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση που διερευνάται αυτόν ε, τον καιρό και σε λίγο καιρό θα δημοσιευτεί η ανεξάρτητη έκθεση της WADA όσον αφορά την διαφθορά στον αθλητισμό στη Ρωσία. Όποιος έχει ασχοληθεί με το θέμα ξέρει ότι οι άνθρωποι που έχουν πάρει μετάλλια στα παγκόσμια πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου η Ρωσία ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη ως προς τα επιτεύγματά της τα τελευταία χρόνια. Φέτος όχι πια, ακριβώς γιατί τους κυνηγάνε. Αλλά πάντως το 12 κέρδισαν περισσότερα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες από τη ΣΥΠΑ. Γίνεται λοιπόν έρευνα, υπάρχει πληροφοριοδότης που μας έχει δώσει ενδείξεις πρωτοφανής και όλες οι ενδείξεις κατατείνουν στο γεγονός ότι οι αθλητές παροτρύνθηκαν από τους ε, ε, προπονητές τους και από τις υπηρεσίες αντι-doping των χωρών τους, της χώρας τους, ότι αν είσαι αρκετά καλός μπορείς και να παραβιάζεις τους κανόνες. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να σταλεί μήνυμα στον κόσμο που θα λέει ότι αν είσαι χώρα που το κάνεις αυτό θα αποκλειστείς για συγκεκριμένα χρόνια. Όχι απλά τους αθλητές, ολόκληρη τη χώρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να αποκλειστεί η Ρωσία. Αν θέλουμε την ευγενή άμυλα πρέπει να της πούμε δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα και να περιμένεις να συνεχίζεις να ε, συμμετέχεις ε, στην, ε, στις αθλητικές διοργανώσεις. Πρόεδρο τη Γουάντα έχει οριστεί από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή δεν έχει συμφέρον από το να μην συμμετέχει η Ρωσία από τους ε, Ολυμπιακούς Αγώνες ε, που θα γίνουν του χρόνου. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί η υπόθεση. Πάντω, αυτό που έχουμε μάθει και έχω μάθει εγώ στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία αυτά τα 37 χρόνια είναι ότι ο αθλητισμό είναι μια όμορφη δραστηριότητα. Είναι ένα όμορφο κόσμο. Αυτό που είπε και η Τζούλι Βόρτ για το χορό. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολείται ένα παιδί με τον αθλητισμό αν ασχολείται ήδη με τον ε, χορό. Τραμπολίνα, ό,τι θέλετε. Αρκεί τα παιδιά να αθλούνται, να έχουν φυσική δραστηριότητα. Αυτό τον τρόπο ζωής θα πρέπει να ε, προωθήσουμε. Τα στοιχεία λένε πολλά. Δεν αρκούν οι Ολυμπιακοί αγώνες να του αναλάβει μια χώρα για να ξεκινήσουν τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Έγινε και στο Λονδίνο αυτό και γίνεται σε κάθε, κάθε φορά που διοργανώνονται Ολυμπιακοί αγώνες. Αν δείτε τώρα το τοπίο και είπατε κι εσείς για τους δύο Ιταλούς που βρέθηκαν, ταινίστες που βρέθηκαν στο US Open αυτό που θέλω να πω είναι αυτοί οι δύο ταινίστρες θα παροτρύνουν περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με το τέννις και αν ναι θα υπάρξουν περισσότερες ε, διοργανώσεις αθλητικές στην Ιταλία, θα υπάρξουν περισσότερες υποδομές, περισσότερες επενδύσεις στον αθλητισμό. Αμφιβάλλω. Γιατί γνωρίζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ξοδεύτηκαν 10 δισεκατομμύρια για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών. Και ξέρω επίσης ότι τα ποσοστά συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις και αθλητικές δραστηριότητες μειώνονται. Και ειδικά, ιδιαίτερα χαμηλά είναι τα ποσοστά σε ε, περιοχές των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι τα παιδιά δραστήρια και ο αθλητισμός πλέον απευθύνεται τουλάχιστον στη Βρετανία στους πλούσιους και στα μεσαία στρώματα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχει σημασία ποια χώρα κερδίζει στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα βελτιώσουμε τα, την καθημερινή ζωή των παιδιών. Υπάρχουν πάρα πολλές διαστάσεις που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον τομέα του αθλητισμού. Δεν μπορούμε να, το, να τα λύσουμε όλα βεβαίως, αλλά χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία. Και αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι αυτό που γίνεται σε επίπεδο πρωταθλητών δεν έχει σημασία. Αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτό που θα πρέπει να, να μας απασχολεί είναι ο μαζικός αθλητισμός και χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους με φυσική δραστηριότητα και θα ήθελα το μήνυμα της σημερινή μου παρέμβασης να είναι αυτό. Χρειάζεται να νομοθετήσουμε για τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό, γιατί εκεί δεν έχουμε κάνει αυτά που πρέπει. Και αν δεν αλλάξουμε ριζοσπαστικά αυτήν την κατάσταση, δεν ξέρω πώς θα αλλάξει συνολικά η κατάσταση. Uh, Σας κατευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Βόλς. Ε, πρόκειτο για την κατάθεσή σας που είναι κάτι ε, σκληρό, αποτελεσματικό, αυτό το οποίο χρειαζόταν να ακουστεί. Ε, αυτό πρέπει να κάνει κανείς, να βάζει ψηλά τον πύχη. Απλώς, ε, πριν δώσουμε το λόγο στους αδέλφους, να πούμε ότι όντως οι Ολυμπιακοί και οι μεγάλες διοργανώσεις δεν βοηθούν για τον κόσμο να σπάσει περισσότερο τον αθλητισμό. Πρώτα πρώτα το θέμα είναι αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε, την άμεση εμπειρία που έχουμε με τα παιδιά, να εμπλέκονται σε αυτές μέσα από την πολιτική. Ε, Επίση να δούμε τι εικόνα προβάλλουμε για τον αθλητισμό. Οπότε η εικόνα κάποιων τίμιων αθλητών είναι πολύ σημαντικό. Σε όλα τα σπορ ε, μπορεί να βρει κανείς και επίσης, όπως είπαμε πριν, για την ποινικοποίηση ε, της ντόπας και του ντοπάζηματος σε όλη την Ευρώπη είναι κάτι βασικό και δεν γιατί κάποιοι διστάζουν να θεσπίσουν το, το αξιόπινο τέτοιων πράξεων. Οπότε έτσι θα πάνε γίνει στην Ευρώπη, πώς θα γίνει να κινηθούμε. Συνάδελφοι και κατόπιν μιλήσουν οι μας. Κυρία Γουόρντ. Ευχαριστώ για την προσέλευσή σας και που μας είπα την προσωπική σας ιστορία. Αυτό χρειαζόμαστε ανθρώπους που βρίσκονται σε υπεύθυνε θέσεις, δασκάλους κτλ. Θέλουμε να είναι και άνθρωποι σας ευχαριστούμε λοιπόν γιατί μας είπατε τα προσωπικά σας. Εγώ είμαι Βρετανή, εκπροσωπώ το βορειοανατολικό τμήμα της Αγγλίας, το βορειοδυτικό τμήμα της Αγγλίας. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ενδιαφερθούμε για πραγματικά προβλήματα incoherent Για τα δίκαια προβλήματα, προβλήματα δικαιοσύνης. Αυτό ψάχνουν και οι πολίτες από τους ηγέτες των... Το ότι ήρθατε λοιπόν εδώ και εκπροσωπήσατε αυτό που εκπροσωπήσατε μου άρεσε πολύ. Καλά, τώρα θα ακούσουμε τους άλλους δύο. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον δεύτερο σύγκρι μας. Ο καθηγητής Ιαν Χένρι από το Πανεπιστήμιο του Λάφμπορο. Ο ρόλος του αθλητισμού για μια ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. see, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ο κύριος. Henry, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας για να κάνουμε αυτή την σύντομη παρουσίαση και να συμμετάσχω και εγώ στη σημερινή σας εκδήλωση. Βέβαια δεν θα το πούμε όλο γιατί υπάρχει χρονικός περιορισμός. Λέμε λοιπόν εδώ ότι βοηθάει ο αθλητισμός στο να χωνέψει κανείς τις διαφορές και να καταπονήσει τις προκαταλήψεις, τον αποκλεισμό, ε, για η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και για ακριβώ τις θετικές συνέπειες του αθλητισμού, αλλά επίσης πολλές φορές έχουμε και κάποιες επικρίσεις. Πρώτα-πρώτα ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για αυτό το οποίο ε, προβάλλεται. Και ε, πολλές φορές έχουμε σεξισμό, έχουμε ξενοφοβία, ε, οπότε και ρατσισμό. Για να δούμε επομένως ε, πώς προάγεται η διαφορετικότητα ε, να δούμε έχουμε εδώ πέρα τρεις διαφορετικές ενότητες που θα σας αναπτύξω. Πρώτα πρώτα το πώς ε, κάποιος αντιλαμβάνεται ε, την ε, πολυπολιτισμικότητα, την εθνικότητα, την ιδιότητα του πολίτη. Δεύτερον, τι γίνεται με το πώς οι ε, τοπικοί παράγοντες προαγάγουν τον αθλητισμό και τρίτον τι στοιχεία υπάρχουν ότι η επαφή μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων μειώνει τις εντάσεις. Πρώτα-πρώτα, επομένως, αυτό το ζήτημα φαίνεται αυτονόητο, αλλά ίσως θα πρέπει να επαναλάβουμε το ότι δεν είναι τόσο ε, ακριβές το ότι όλα τα σπορ είναι καλά για όλους. για τον καθένα κάτι άλλο είναι πιο ωφέλιμο, διαφορετικό σπορ. Να δούμε λοιπόν ποιος ωφελείται από ποιο σπορ. Οπότε το πρώτο μας θέμα τώρα είναι η σχέση μεταξύ πολυπολιτισμικότητας, διαπολιτισμικότητας, ιδιότητας του πολίτη και προσέγγιση στην ε, πολιτική του αθλητισμού. Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες όσον αφορά την ένταξη, όσον αφορά την αφομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το πώς το ένα αντιτίθεται στο άλλο. Είναι θέματα εθνικής ε, ταυτότητας, ιδιότητας του πολίτη, δικαιώματα του πολίτη. Οπότε, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα κλασικό πλαίσιο για τις πολιτικές που θα χρησιμοποιήσουν για την κοινωνική ένταξη τον αθλητισμό, θα έλεγα ότι έχουμε τρία ε, πρότυπα, τρία κλασικά μοντέλα. Πρώτα-πρώτα, το γαλλικό μοντέλο όλοι δηλαδή οι πολίτες της Γαλλικής Δημοκρατίας να μπορούν να έχουν αθλητισμό και η θρησκεία και οι πολιτισμικές προτιμήσεις περνάνε στο ιδιωτική σφαίρα της ε, δημοκρατίας. Δεύτερον έχουμε το γερμανικό μοντέλο. Υπάρχει και ιδιωτική διάστημα στο γαλλικό μοντέλο αλλά στο γερμανικό μοντέλο ε, έχουμε τα δικαιώματα από το πολιτικό όραμα το οποίο αφορά τον αθλητισμό. Επίσης έχουμε το αγγλικό πρότυπο το οποίο έχει να κάνει και με το αποκυκρατικό παρελθόν της Βρετανίας. Βεβαίως αυτά όλα τα μοντέλα αλλάζουμε το χρόνο αλλά υπάρχουν κάποιες σταθερές οπότε έτσι μπορούμε εμείς να τα δανειστούμε για να δούμε τι πλαίσιο πολιτικής θα φτιάξουμε. Τώρα για να δούμε εδώ έχουμε έξι διαφορετικά μοντέλα. Πρώτα πρώτα διαπολιτισμικότητα ε, κοινωνική νοοτροπία και κατόπιν έχουμε μέσω του αθλητισμού επομένως την χρηματοδότηση, υποστήριξη του πολιτισμού. Δεύτερον, έχουμε όλες τις πολιτιστικές ε, υπηρεσίες της κλασικής δημοκρατίας, ισότητα ευκαιριών και εδώ έχουμε επίσης την χρηματοδότηση πολιτιστικών ανταλλαγών. Επομένω, η κατάληξη αυτή τη προσπάθεια είναι η προσβασιμότητα από όλου στον αθλητισμό. Μετά έχουμε την πιο επίμαχη αρχή της προσέγγισης από πλευράς ε, γαλλικής νοοτροπίας γιατί από πλευράς πολιτικής η προστασία των πολιτικών μειονοτήτων ας πούμε ε, να έχουμε κάποιες ε, έδρες στο κοινοβούλιο για κάποιες ομάδες ε, αποσκοπής, στο να προστατεύσουμε κάποιες αδύναμες πολιτικές, κοινωνικές ε, ομάδες. Και επίσης ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει μέσω των συλλόγων και των εκδηλώσεων. Τέταρτον, έχουμε την πολυμορφία της αγοράς, τον πλουραλισμό της αγοράς. Ας πούμε οι μουσουλμάνες να μπορούν να αθληθούν και να μπορούν να πάνε στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Έχουμε εδώ τη συγκερασμό του εθελοντισμού με την εμπορικοποίηση. Μετά έχουμε το πώς μπορεί να έχουμε κάποιο είδους αφομοίωση αυτών των πολιτικών. Εδώ είναι το εύκολο σύστημα. Γιατί μπορούμε να θεωρήσουμε εδώ ότι είναι όχημα ο αθλητισμός για να προσδώσει κάποιου κοινωνικά ωφελήματα και να μην στοχεύει συγκεκριμένες μειονότητες. Αυτό αφορά συνήθως ομοιογενείς πολιτισμούς και γίνεται με τις αντίστοιχες πολιτικές. Βλέπετε εδώ όλο το φάσμα των προσεγγίσεων που υπάρχει. Κατά τον τρόπο Αυτές όλες οι πολιτικές στηρίζονται σε διαφορετική κατανόηση, διαφορετικές προσδοκίες για το τι ωφελήματα μπορεί να προκύψουν από την παρέμβαση μέσω του αθλητισμού. Επομένως, τι ισχύει όσον αφορά τα ωφέλη και από αυτούς που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών αλλά και εκείνους οι οποίοι ε, εργάζονται για τους προηγούμενους στη βάση. Έχουμε εδώ το θέμα των προσφύγων, των ετούντων άσυλο, στα κέντρα υποδοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο και μπορώ να σας δώσω τρία παραδείγματα. Για κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μας βοηθήσουν να αντιλήσουμε συμπεράσματα. Πρώτα-πρώτα είναι η κοινότητα Βοσνίων στο Ντέρμπι. Εκεί αμέσως μετά τον εμφύλιο στην Κυκλοσλαβία ξεκίνησε αυτή η εγκατάστασή τους και εδώ έχουμε αυτό το success story. Γιατί οι εκεί οι Βόσνοι μπόρεσαν να συνεργαστούν με τους υπολείπους όσον αφορά το μπασκετμπόλ γιατί είχαν δεξιότητες καλύτερες από ότι οι Βρετανοί οπότε είχαμε ανταλλαγή παικτών και έτσι είχαμε στενές σχέσεις μεταξύ Βοσνίων ε, και Βρετανών που παίζουν στο πρωτάθλημα. Εδώ τα δείχνει βέβαια όλα ρόδινα γιατί είναι αυτό το οποίο έγινε στην αρχή μόνο, στην αρχή. Αλλά βλέπουμε ένα παράδειγμα του πώς μπορεί κανείς να αποσπάσει κάποια ωφέλη. Δεύτερο παράδειγμα είναι κάτι που έχει να κάνει με τους Κούρδους πρόσφυγες. Και αυτοί στην ίδια πόλη, στον Τάρμπι, η συσχέτισή τους με διάφορους μουσουλμάνους, με Βρετανούς Πακιστανής καταγωγής κλπ. Εδώ είδαμε ότι είχαμε τις υπηρεσίες κοινωνική πρόνοιας, είχαμε την αστυνομία και όλοι συνεργάστηκαν ούτω ώστε να ιδρυθούν κάποιοι αθλητικοί σύλλογοι όπου θα συμμετείχαν και οι μεν κοινότητες και οι δε κατά της ε, βίας οπότε χρησιμοποιήθηκε δηλαδή αυτού του είδους ε, ε, η πρωτοβουλία του αθλητισμού το ώστε να έχουμε συνεργασία και κάλυψη των ατομών αυτών στην παιδεία, στη στέγαση κλπ. Αλλά βλέπουμε πως το κεφάλαιο του αθλητισμού αξιοποιείται σε άλλους τομείς. Τρίτο παράδειγμα. η αλγερινή στο Νότιγχαμ. Δεν ήταν μόνο αλγερινή ήταν από όλη την Αφρική. Εδώ υπήρχαν ορισμένε υπηρεσίες που απίλαυναν ε, μείναν κάπως κλειστοί και ε, συνεργάστηκαν μόνο με όποιους είχαν παρόμοιες ε, εμπειρίες, τραυματικές εμπειρίες ε, σαν τον άσυλο ή σαν πρόσφυγες. Οπότε έχουμε εδώ τρία διαφορετικά είδη κεφαλαίου αθλητικού. Και όταν μιλούσαμε με αυτά τα πρόσωπα, γιατί έτσι έγινε αυτή η μελέτη από τη βάση, αυτοί που ζουν εκεί, που είναι αποδεκτών των υπηρεσιών που είπαμε, ανέφεραν προσωπικό όφελος σε επίπεδο υγείας, ψυχολογικής υγείας, όσον αφορά τις, το, στρες, την ένταση ε, της καθημερινής ζωής. Αν και θυμάμαι και έναν Κογκολέζο που έδινε μια συνέντευξη και έλεγε ότι χαμογελά μόνο την Κυριακή. Γιατί τότε πήγαινε στο συγκεκριμένη λέσχη, στον φορέα. Γιατί όλη την εβδομάδα πήγαινε από δουλειά σε δουλειά. Οπότε να βλέπουμε ποια είναι τα προσωπικά ωφέλη. Επίσης, έχουμε ωφέλη από πλευράς κοινωνικής. Είπαμε ότι ο αθλητισμός έγινε γέφυρα Βοσνίων και Βρετανών γιατί οι αθλητές έτσι ε, ήξερε η τοπική κοινωνία πού θα πάει να βρει τους ε, Βόσνιους πρόσφυγες να τους παρέχει ό,τι υπηρεσίε παρήχονται γιατί και τους ήξερε από τον Αθλητικό Σύλλογο. Άρα εδώ πέρα είχαμε προσέγγιση, είχαμε αυτή την προϋπόθεση για την υποστήριξη ε, αυτών που κατά τα άλλα ήταν ε, ανήμποροι. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό έχει να κάνει με τους, τα δύο διαφορετικά είδη και στόχους Πολιτική που είπαμε στην αρχή. Και έχουμε αυτά τα στοιχεία για το πώς μπορεί να υπάρξει κάποιο όφελος σε μικρή κλίμακα για τους ε, πρόσφυγες. Αλλά, αλλά σε μεγάλη κλίμακα τι γίνεται. Μας πείθουν τα στοιχεία που έχουμε ότι η επαφή μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων μειώνει τι εντάσει. Νομίζω ότι σημειώσαμε μια πραγματική επιτυχία για την ποιότητα των στοιχείων. Και πετύχαμε γιατί είχαμε νέους τρόπους συλλογή των στοιχείων. Και έτσι είδαμε την ευρύτερη εικόνα, το ευρύτερο τοπίο. Θα σας πω ποιες ήταν οι πηγές των στοιχείων. Πρώτα-πρώτα. Είχαμε την μελέτη πολλών υποθέσεων από το αρμόδιο Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού και μια βασική πηγή ήταν αυτή η συστηματική μελέτη που έγινε με 232 επιμέρους μελέτες. Και έτσι εκμεταλλευθήκαμε το αθλητικό κεφάλαιο από αυτές τις αθλητικές πρωτοβουλίες, οπότε από όλες αυτές τις μελέτες αντιλήσαμε αδιάσυστα στοιχεία. Αλλά ακόμα πιο ενθαρρυντικό ήταν αυτού του είδους η συλλογή στοιχείων. Αυτή η μεταανάλυση, 515 εμπειρικές μελέτες, από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα. Και αυτές οι μελέτες έγιναν σε 25 χώρες. Όχι μόνο για αθλητισμό, αλλά και για πολιτισμό, για παιδεία κλπ. Πάρα πολλοί τομείς. Καλύφθηκαν όπου υπάρχει διαπολιτιστική επαφή κοινωνικών ομάδων. Τα στοιχεία είναι διάστητα. 94% ε, των ε, ερευνών είναι θετικών συμπερασμάτων. Πρόκειται για επιχειρήματα τρανταχτά, διάσυστα που προκύπτουν. Το δε υλικό που συνελέγει από τη δεκαετία του 50 για την ε, θεωρία της επαφής των πολιτικών ομάδων ξεκίνησε από έναν ε, Αμερικανό επιστήμονα. Και τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς επιχείρηματα κατά αυτής της θεωρίας. Να, βλέπετε κάποια παράδειγμα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο αθλητισμός ε, στα πλαίσια αυτών των 515 ερευνών. Πέραν αυτών, μπορέσαμε να δούμε σε ποιε συνθήκες η επαφή των ομάδων γίνεται πιο αποτελεσματικά να υπάρχει, να υπάρχει ισότητα των ομάδων, να υπάρχει συνεργασία, ε, ανταγωνισμός για επίτευξη κοινών στόχων, ε, σεβασμός προς κάποιες αρχές που να στηρίζουν, οπότε αυτή η συνεργασία θα πρέπει να γίνεται ε, σε προσωπικό επίπεδο και όχι έτσι απλώς τυπικά σε επίπεδο κοινότητας κλπ. Οπότε τώρα βλέπετε ότι έχουμε αυτά τα σειρά επιχειρήματα κατά των κοινικών Επίση έχουμε και κάποιο είδους γενικόλογες, γενικού χαρακτήρα προποθέσει επιτυχίας, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά στον πολιτισμό και σε άλλους τομείς. Οπότε βλέπετε ότι έχουμε κάποια στιγμή που είχαμε πριν και έχουμε κάποιου πανεπιστημιακού συναδέλφου, οι οποίοι μπορεί να είναι αρνητικοί ε, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι πανεπιστημιακή παράδοση όταν κάνει αντιρρησίας. Τέλος πάντων. Okay. So, Λοιπόν, σαν συμπέρασμα. Δεν θα σας διαβάσω όλα, αλλά αυτό που ελπίζω ότι σας όταν καταλάβετε είναι μια σύνοψη αυτής μου της εργασίας. Είναι δηλαδή μια αισιόδοξη άποψη της χρήσης του αθλητισμού, για την επαφή διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, να έχουμε που προκαταλήψει και έτσι να υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ αυτών των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη που αναφέρατε και τα πρότυπα. Α, πάρα πολύ ωραία. Και τα θετικά συμπεράσματα που αναφέρατε. Ευχαριστούμε και θα δώσουμε τον λόγο στην ε, επομένη εισηγήτρια. είναι η δόκτωρ Άννα Κλάισνερ. Αφορά την οικονομική διάσταση του αθλητισμού. Νέο θέμα και ενδιαφέρον. Γιατί πριν μίλησα με τον Υπουργό και μίλαγαμε για την οικονομική βιωσιμότητα του αθλητισμού. Είναι θέμα που θα απασχολήσει εις βάθος την Λουξεμβουργενή Προεδρία δουλεύετε για το Υπουργείο Αθλητισμού της ε, Αυστρίας και για το αντίστοιχο ε, αθλητικό ίδρυμα. Έχετε και εσείς 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και χαίρομαι που θα σας μιλήσω για την οικονομική διάσταση του αθλητισμού. Θα σας πω και ποια είμαι. Λέγομαι Άννα Κλάσνερ και είμαι ανώτατη ερευνήτρια στο Ίδρυμα για τον Αθλητισμό της Βιέννης που στοχεύει στην ποσοστικοποίηση των στοιχείων για τον αθλητισμό και προμηθεύει στατιστικά στοιχεία και σε άλλες χώρες. Θα μπορούσα να σας μιλήσω δύο ώρες για την οικονομική διάσταση του αθλητισμού, αλλά σε μόνο 15 λεπτά πρέπει να περιοριστώ. Στα κυριότερα. Θα σας μιλήσω λοιπόν πρώτον για τον οικονομικό ορισμό του αθλητισμού. Γιατί αν και φαίνεται σαφής είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί. Μετά α, γενικότερα για την οικονομική επίπτωση του αθλητισμού, μακροοικονομικές επιπτώσεις και αριθμούς στο ΑΕΠ ή στην απασχόληση. Μετά μερικές λεπτομέρειες για τις εθνικές αδυναμίες ή ωφέλη μεταξύ χωρών και τις δυνατότητες που έχουν. Αν σκεφτούμε τον αθλητισμό στην Ευρώπη, καταλαβαίνουμε εύκολα ότι έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Συμμετέχει στην ανάπτυξη αυξάνει το ΑΕΠ, δημιουργούνται θέσεις εργασίας και άλλα. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν 0,8% ε, ε, και 0,3% στο ΑΕΠ 0,8 και 0,3 στην απασχόληση. Αυτό φαίνεται να είναι αντιφατικό. Υπάρχουν λόγοι όμως για αυτή τη διαφορά. Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις του αθλητισμού έχουν υποτιμηθεί γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ του στατιστικού εύρου των στοιχείων και της κοινή αντίληψης για τον αθλητισμό. Δηλαδή, έχουν λάβει υπόψη τους κυρίως αθλητικές οργανώσεις και εγκαταστάσεις, οργανωμένες λέσχες κλπ. Αλλά υπάρχουν αθλητικές δραστηριότητες και σε άλλους τομείς, σε επιχειρήσεις, στον τουρισμό και για πολύ καιρό δεν υπήρχε επίσημος ορισμός του αθλητισμού. Από το 7 όμως έχουμε. Πριν δεν ήταν δυνατόν να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μελετών μεταξύ χωρών και γενικά δεν υπήρχαν πολλά στοιχεία συγκρίσιμα. Ούτε γνωρίζαμε τις λεπτομέρειες για τους υποτομείς του αθλητισμού και δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια ποσοτική ανάλυση σωστή. Τώρα έχουμε τον, την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον αθλητισμό και τη στατιστική. Θα αρχίσω με τον ορισμό του αθλητικού τομέα. Η εικόνα εδώ που βλέπετε είναι μια απλοποιημένη περιγραφή του θέματος. Δείχνει τις πολλές επιπτώσεις που έχει ο αθλητισμός επί της οικονομίας. Το πρόβλημα είναι ότι Μόνον αν υπάρχει σαφής ορισμός του τι τομείς και υποτομείς συμπεριλαμβάνονται, μόνο τότε μπορούμε να μετρήσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις. Εμείς είδαμε ότι δεν είναι χρήσιμος ένας και μόνο ορισμός. Ε, γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε έναν τριπλό. Το στατιστικό ορισμό, δηλαδή τη λειτουργία του οργανωμένου αθλητισμού με λέσχες κλπ. Μετά αν προσθέσουμε και τους υπόλοιπους τομείς που ενδιαφέρουν τον αθλητισμό, που χορηγούν υπηρεσίες κλπ. Τότε έχουμε τον στενό ορισμό, παραδείγματος χάρη, για να παίξει κανείς ποδόσφαιρο χρειάζεται μπάλα, ρούχα, παπούτσια, στάδιο κλπ. Στον ευρύ ορισμό έχουμε όλους τους άλλους τομείς που κάπως συνδέονται με τον αθλητισμό αλλά δεν είναι απαραίτητη για να υπάρξει ο αθλητισμός ας πούμε, οι αθλητικές ειδήσει και τέτοια. Αυτός ο τριπλός ορισμός λοιπόν χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στην Αυστρία από το 7. Η μέθοδοι μετρήσεως του αθλητισμού είναι μέσω ενός ειδικού συστήματος που δεν είναι απεσήμως τμήμα των εθνικών λογαριασμών για τη συμβατότητα με άλλα εθνικά συστήματα είναι απαραίτητη η συμβατότητα αυτή αν θέλουμε να συγκρίνουμε αλλά και να κάνουμε συγκρίσεις με άλλους μακροοικονομικούς ή μικροοικονομικούς υποτομείς του αθλητισμού. Είναι βέβαια πολύπλοκη και ακριβή διαδικασία, το είδαμε αυτό στην πράξη, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε την εργασία αυτή γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να μετρήσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις. Πώς γίνεται λοιπόν, αυτή, πώς εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος, δεν είναι δύσκολο. Παίρνουμε τα εθνικούς πίνακες input-output, τους μοιράζουμε σε σχετικούς ή άσχετους με τον αθλητισμό και τελικά τους συνδυάζουμε και τα συνδυάζουμε τους εθνικούς πίνακες και έχουμε μία πανενοσιακή σύγκριση, ένα πανενοσιακό πίνακα. Uh, Ακούγεται απλό γιατί αρχίζουμε από απλούς πίνακες input-output αλλά εδώ βλέπετε στις στήλε ας πούμε τι προϊόντα πολλούνται στην ενδιάμεση κατανάλωση και στην τελική κατανάλωση στις στήλε δε βλέπετε επίσης τι άλλο πρέπει να παραχθεί για να υπάρξει αθλητισμός. Στην 27 χώρες μέλη και άρα 27 πίνακες input-output. που έπρεπε να συνδυάσουμε. Ο κάθε τομέας που σχετίζεται με τον αθλητισμό υποδιαιρείται και ό,τι αφορά τον αθλητισμό το βάζουμε σε χωριστή στήλη. Για τις 27 χώρες το κάναμε αυτό και τελικά έπρεπε αυτούς τους 27 πίνακες να τους συνδυάσουμε για να έχουμε έναν ενωσιακό πίνακα input output. Άμα δούμε μόνο το κεντρικό τμήμα τότε έχουμε 27 περιφέρειες με 94 υποτομής 2.538 δηλαδή κυψέλες. Άρα είναι δύσκολα, δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Εδώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω ορισμένα αποτελέσματα της μελέτης μας. Καταρχήν τον ευρύ ορισμό του αθλητισμού που, με τον οποίο φαίνεται ότι 1,7 προστιθέμενης αξίας οφείλεται στην Ευρώπη στον αθλητισμό. Ε, άμεσα. Με απόλυτους όρους ο αθλητισμός ευθύνεται για 173 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οι έμεσες επιπτώσεις τώρα φτάνουν σχεδόν στο 3% support on the European level is therefore comparable to the agriculture, forestry and fishing sector. Ενώ και τα λοιπά. Οι σημαντικότεροι τομείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό είναι οι βοηθητικές υπηρεσίες, οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, οι υγειονομικές υπηρεσίες και η λιανική. Είναι σημαντικό, φαίνεται εδώ πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε το πραγματικό ορισμό της επιπτώσεις στην απασχόληση ας πούμε σύμφωνα με τις, τα τρία τμήματα του ορισμού 0,3% μόνο στο στατιστικό σκέλος αλλά 2% στον ευρύτερο και παραπάνω από 2% για την απασχόληση. 1,76% και άρα ο αθλητισμός ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την απασχόληση. Εδώ βλέπετε μερικές λεπτομέρειες εθνικών πινάκων. Γενικά στην Ευρώπη συνολικά έχουμε 4,5 εκατομμύρια ανθρώπους που απασχολούνται άμεσα με τον αθλητισμό, στον αθλητισμό. Η ψηλότερη ρυθμή στην Αυστρία και το Λουξεμβούργο σε σχετικούς αριθμούς όμως. Τώρα οι αδυναμίες ορισμένων χωρών προσπαθήσαμε να βάλουμε μία βαθμολόγηση από 1 μέχρι 27 ανάλογα με την αθλητική παραγωγή τα κύρια αποτελέσματα βρίσκονται εδώ, εδώ. Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Αυστρία και Πολωνία έχουν πολύ ψηλό βαθμό. Γερμανία επίσης στις υπηρεσίες και στα αγαθά η Σλοβενία σχεδόν σαν τη Γερμανία στα αγαθά, αλλά όχι τόσο πολύ στις υπηρεσίες. We were looking at Τώρα οι αναπτυξιακές δυνατότητες σχεδόν σε όλες τις χώρες τρεις τομείς είναι πολύ υποσχόμενοι η αθλητική διατροφή, οι αθλητικές ασφαλίσεις. και η χορήγηση νομικών συμβουλών. Ο πολλαπλασιαστής δηλαδή είναι τουλάχιστον δύο. δύο. Τώρα οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ χωρών. Στις ομοιότητες οι χώρες με το μεγαλύτερο ΑΕΠ κατά ανακεφαλή έχουν και υψηλότερο μερίδιο στις αθλητικές δραστηριότητες. Όχι μόνο σε απόλυτους αλλά και σε σχετικούς αριθμούς. Σε όλες τις χώρες έχουμε τους τρεις υποσχόμενους τομείς που σας ανέφερα πριν και οι υποβοηθητικές υπηρεσίες στις μεταφορές όπως οι ταξιδιωτικές ε, υπηρεσίες κτλ. Οι διαφορές τώρα μεταξύ των χωρών δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε όλες τις χώρες. εμένα είναι εύκολο να αναφερθώ στην Αυστρία γιατί είναι από τις κυριότερες χώρες στον αθλητισμό και υπάρχει λόγος γι' αυτό γιατί τη χειμερινή περίοδο έχουμε βουνά και γίνεται σκι και μεγάλο τμήμα του αθλητισμού σχετίζεται με τον τουρισμό ενώ αντίθετα στην Κύπρο τα κύρια αθλητικά γεγονότα είναι από μακριά. Η Γερμανία έχει πολύ μεγάλη ιδιωτική κατανάλωση αθλητισμού. Κατανάλωση. Κάτι παρόμοιο για την Ολλανδία. Ίσως Ηνωμένο Βασίλειο να ήταν ενδιαφέρον επίσης. Γιατί η κατανάλωση που σχετίζεται με τον αθλητισμό επλήγει δυστυχώς από την κρίση. Αλλά η ολυμπιακή του Λονδίνου όθησαν τα πράγματα και γι' αυτό φτάσαμε στα ίδια. Μπορώ να τελειώσω εδώ αν θέλετε και σας κατευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. Σας ευχαριστούμε λέει η Πρόεδρος. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας. Σίγουρα θα εμβαθύνουμε από τις ε, σίγουρες ερωτήσεις που έχουν να υποβάλουν οι συνάδελφοι. Και τώρα να δώσουμε τον ε, λόγο στον ε, κύριο Λοστέκ για το θέμα αθλητισμός και ισορροπία στη ζωή. Μήπως πριν δώσουμε το λόγο στον επόμενο μιλή μας έχει να κάνετε κάποιες ε, ερωτήσεις αν δεν έχετε να ολοκληρώσουμε με αυτή την ομιλία και αν συμφωνείτε ρωτάτε μετά έχουμε και τον κύριο Φίζας ο οποίος ε, αναφέρθηκε τόσες φορές μια που ήταν ο συντάκτης της έκθεσης του Κοινοβουλίου για τον αθλητισμό. Οπότε να ολοκληρώσουμε και κατόπιν θα δώσω λόγο συναδέλφια. Merci, merci beaucoup, Madame. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την πρωτοβουλία σας να οργανώσετε αυτό το σημαντικό σεμινάριο. Είναι σίγουρα καυτό το θέμα. Ο αθλητισμός όλο ένα και περισσότερο ε, αναγνωρίζεται για τη σημαντική θέση που έχει στη ζωή όλων μας. Είναι πολύ σημαντική συγκυρία γιατί ολοκληρώνουμε την πρώτη ε, ευρωπαϊκή βδομάδα αθλητισμού στις Βρυξέλλες διάλογος συνεχίζεται. Οπότε να, είναι σωστή ώρα να τα πούμε για αυτό το σημαντικό θέμα. Οπότε, πρώτα-πρώτα δύο λόγια προσαγωγικά. Ας κάνουμε ένα βήματάκι προς τα πίσω. Το 2014 νομίζω ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον αθλητισμό όσον αφορά την, ε, ε, τις επιδόσεις μας για επιτροπή, για συμβούλιο, για κοινοβούλιο γίνανε σημαντικά πράγματα. Το 2014 ήταν το πρώτο έτος ε, υλοποίησης του Έρασμος ΣΥΝ, το πρόγραμμα το οποίο επιψηφίσατε η πρώτη χρονιά της υλοποίησης της σύστασης του Συμβουλίου για την ε, προώθηση της ε, σωματικής δραστηριότητας. Επίσης τότε εγκρίθηκε το δεύτερο πρόγραμμα εργασίας 14-17 και είχαμε πρώτη φορά που περιλήφθη στο χαρτοφυλάκιο ε, επιτρόπου ο αθλητισμός. Επομένως το 2014 ήταν μια καλή χρονιά και το 2015 όμως ξεκίνησε ε, το ίδιο καλά, αν όχι καλύτερα, γιατί το 2015, ε, όπως θα δούμε σε λίγο, είχαμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα του Αθλητισμού. Είχαμε επίσης αυτές τις ε, επαφές και συζητήσεις για τους ΣΥΚΕ αγώνες. Αυτό νομίζω ότι θα μας οδηγήσει σε πρόοδο. Επίσης, είχαμε και έναν προβληματισμό στους κόλπους της Επιτροπής σε συνεργασία με τα κρατημέλη, αλλά και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο όσον αφορά τον επαναπροσανατολισμό του έρασμος συν ούτως ώστε να καλύψουμε περισσότερο ε, το σπορ ε, στη βάση της κοινωνίας. Επομένως όλα αυτά τα ωραία γίνουν το 15. Και τώρα, μια που μιλούμε για τον λαϊκό αθλητισμό, με το λαϊκό στη βάση, ερχόμαστε στο θέμα μας. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Γενικώ την προώθηση της σωματικής ε, δραστηριότητα. Να δούμε ποιος είναι ο στόχος. Είναι πάρα πολύ απλός. Με μια φράση το τον εκφράζουμε. Να αυξηθεί η συμμετοχή στον αθλητισμό και την σωματική δραστηριότητα. Ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνούμε όμως ότι η δραστηριότητα δεν πάει να πει να είναι κανείς γραμμένος σε αθλητικό σύλλογο. Ξέρετε επίσης ότι είχαμε διάφορα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο και λέει ότι 41% των Ευρωπαίων κάνουν ε, αθλητισμό λίγο ή καθόλου δεν κάνουν. Και αυτό είναι πίσω γύριμα σε σχέση με άλλη προηγούμενη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του 2009. Γιατί μεταξύ 9 και 14 αυτοί που δεν κάνουν ποτέ αθλητισμό από το 39% πήγε στο 42%. Επομένως αυτό είναι κακά μαντάτα. Ακριβώς ε, αυτές οι πρωτοβουλίες αυτό θέλουμε να κάνουν. να αντιμετωπίσουν τέτοιες προκλήσεις τώρα. Όσον αφορά τους στόχους για να μπορούμε το τοπίο να το συμπληρώσουμε. Κάποιος, έλαβε το λόγο πριν και είπε ότι βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να τα κάνει όλα μόνη της με τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει το λιθαράκι της αλλά γνωρίζει ότι οι εταίροι της κρατούν το κλειδί. Τα κρατεί μέλη, οι κρατικές αρχές, οι κοινοτικές αρχές, οι ομοσπονδίες και σύλλογοι οι αθλητικοί. Άρα βλέπετε ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι ταπεινός ο ρόλος μας, αλλά θα πρέπει αυτό το ρόλο τέλος πάντων να τον αναπτύξουμε σε συνεργασία με τους άλλους. Τώρα, δύο λόγια για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Δεν είναι αυτός σκοπός. Ο στόχος είναι να γίνει δουλειά μακροπρόθεσμα για να προωθηθεί η δραστηριότητα, ο αθλητισμός και έτσι να έχουμε μια μακρόπνοη πολιτική. Να μην επεκταθώ πάνω σε αυτό, αλλά γνωρίζετε ότι έχουμε ένα ε, εργαλείο που εδώ το ψηφίσετε στο το Έρασμος ΣΥΝ όπου κάποια τμήματα του προγράμματος προάγουν ακριβώς σωματική δραστηριότητα, αθλητική δραστηριότητα να, αυτό κάναμε στην ε, εβδομάδα χρηματοδοτήσαμε κάποια προγράμματα κάποια, κάποιες εκδηλώσεις μία εκδηλώση ανά κράτος μέλος με τα περίφημα σημεία συντονισμού, εθνικά σημεία συντονισμού και βλέπετε τώρα πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Το 2015 είχαμε 25% του προϋπολογισμού που πρικοδότησε όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα αλλά και κάποια προγράμματα που αφορούν τη συνέχιση της προσπάθειας το 2015. Ε, λίγο πιο κάτω από το 20%. Το 2016, συγγνώμη, αλλά δεν προσθέθηκαν άλλα λεφτά, οπότε αν και έπεσε το ποσοστό ήταν σημαντικό ότι πήγαμε λίγο παραπάνω από το 20%. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Τι είναι το νόημά της, ποιο είναι το νόημά της, τι πνεύμα της προσδώσαμε, πρώτα πρώτα θα πρέπει να πούμε, πάλι με κάθε μετρή ευρωσύνη, ότι δεν μας ήρθε μας η ιδέα ως επιτοπλίστων ξεπίδησε αυτή η ιδέα από την έκθεση φύσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έπαιξε επομένως σημαντικό ρόλο ο κύριος Φύσας. Οπότε πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου ε, ήταν που μας έδωσε το σπέρμα αυτής της ε, πρωτοβουλίας. Από εκεί πήραμε την ιδέα, οπότε και το Συμβούλιο τελικά ενώσε τι προσπαθίε του, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να μα ανέθεσε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Ξέρετε τις ε, προηγούμενη εβδομάδα στι βρυξελλε 7 7-13 Σεπτεμβρίου, αλλά ένα κλειδί στην επιτυχία της εβδομάδα ήταν η ευελιξία. Το τελευταίο το οποίο ε, θα έκανε η Επιτροπή ήταν να ερχόταν και να έλεγε «Για κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα είναι αυτές τις μερομήνιες και έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Ακριβώς αυτό δεν θέλαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι το να λάβουμε υπόψη όλα τα παραδείγματα προς μίμηση όλων των κρατών μελών, όλες τις επιτυχείς εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε να υπάρξει μια μεγάλη ευελιξία στις εθνικές, περιφερειακές, τοπικές πρωτοβουλίες του αθλητικού κινήματος για αυτήν την εβδομάδα. Και έτσι και έγινε. Επίσης, πηγή έμπνευσης ήταν κάποια κρατημέλη και κάποιοι αθλητικοί φορείς που έκαναν αυτές τις focus days. Κάποιες ημέρες δηλαδή όπου αναπτύχθηκε αθλητική δραστηριότητα ε, στην παιδεία, στο σχολεία, πανεπιστήμια σε επιχειρήσεις, γενικά σε χώρους εργασίας, κάναμε πολλά, αρχίσαμε εντατικά να ε, δουλεύουμε εκεί πέρα, αλλά επίσης και ο αθλητισμός ε, σε υπαίθριους χώρους, outdoor, αλλά μην ξεχνούμε επίσης τα γυμναστήρια, τους αθλητικούς συλλόγους, αλλά και τις ε, αθλητικές ενώσεις που είναι το λίκνο του, του, του αθλητισμού και ας μην έχουν την αποκλειστική δραστηριότητα. Επίσης, έχουμε 10 πρεσβευτές οι οποίοι έχουν ως κοινό σημείο κάτι συγκεκριμένο. Είναι περισσότεροι γνωστοί, άλλοι λιγότερο γνωστοί. Έχουμε δύο πάρα πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές, αλλά επίσης και άλλους που προέρχονται από σπορ λιγότερο γνωστά. Και αυτοί οι πρέσβεις ακριβώ προβάλλουν την εικόνα αυτών που κάνουμε. Δηλαδή είναι κάποιοι που τους αγαπάει ο κόσμος είναι κάποιοι αναγνωρίσιμοι. Άρα και εμείς ε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την επιλογή αυτών που κάνουμε για πρεσβευτέ. Οπότε έτσι μπορέσαμε να προβάλλουμε το έργο μας πολύ. Επίσης έχουμε και την εκστρατεία ενημέρωσης πολύ σημαντική και επικοινωνίας τον Ιούνιο. Επίσης ε, όσον αφορά κάθε αυτή την εκδήλωση της Βρυξέλλες είχαμε πολλούς που ενεπλέκησαν είχαμε τη Δευτέρα την ενακτήρια εκδήλωση, είχαμε την Τετάρτη μια διάσκεψη, όλη εβδομάδα υπήρχε ένα χωριό που τα πήγε πολύ καλά σε μια πλατεία. Όλα αυτά πολύ σημαντικά. Αλλά πιο σημαντικό είναι το τι έγινε σε όλα τα κρατημέλη. Οπότε οι συνεργάτες μας, ε, που και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, ε, ήταν 30 ε, φορείς αθλητικοί, 25 μέτρα ενημέρωση και, ε, και άλλοι φορείς. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά ε, την Ευρωπαϊκή αυτή εβδομάδα, το τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένω όλα αυτά συνέβαιναν σε επιτυχία. Τώρα για την τελευταία διαφάνεια, μια τελευταία λέξη, ότι σε κάθε γλώσσα έχουμε αυτό το εθνικό σημείο κόμβο συντονισμού 33 κράτη-μέλη από αυτά, από τα 33 τέλο πάντων, 31 κράτη-μέλη συμμετέσχουν. Και ένα κρατος κράτος ήθελε πρώτα πρώτα να περιμένει να δει πώς πάνε τα πράγματα και πριν τελικά προσχωρήσει στην προσπάθεια. Θα δούμε. Τώρα δε, τι ανάλυση μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά είναι ακόμα πρώιμο αυτό. Τώρα τελείωσε η πρώτη εβδομάδα, τα εκδηλώσει συνεχίζονται σε κράτη-μέλη, αλλά πάντως όλες οι ενδείξεις ε, είναι ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Είχαμε υποστήριξη πολιτική, πολύ σημαντική, πολύ καλό για μας, γιατί μια τέτοια πρωτοβουλία δεν μπορεί να βαδίσει, να σταθεί μόνη της. κάποια κρατή-μέλη και κάποια νομικά πρόσωπα βοήθησαν με ενθουσιασμό. Επίσης για τις συνεργασίες, είπαμε είχαμε 30 τέτοιους συνεργάτες, μεγάλες τελικέ ομοσπονδίες συνεργάστηκαν για να εξαφανιστεί συνέχεια. 3.000 μέχρι στιγμής εκδηλώσεις, είπαμε σε 31 μέλη. 5 εκατομμύρια συμμετέσχων, οι οποίοι αυξάνονται, αυγατίζουν συνέχεια. Και να δούμε τι θα γίνει σε κάτι Τώρα, για να κλείσω όσον αφορά την συνέχεια για την επόμενη μέρα όλα θα εξαρτηθούν από εμάς όλους εμάς από την Επιτροπή θα κάνουμε μια ανάλυση αλλά και από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Αθλητικές Ομοσπονδίες θα κάτσουμε να αξιολογήσουμε θα προσπαθήσουμε να είναι σοβαρή ενδελεχής η ανάλυση να δούμε πώς τα πήγε σε κάθε περίσταση αυτή η πρωτοβουλία. Και σε Σεπτέμβριο του 2016 θα έχουμε τη νέα προσπάθεια και το τι θα γίνει θα εξαρτηθεί από το τι θα πει ο καθένας ε, όπου συζητηθεί αυτή η αξιολόγηση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πρόεδρος για τις τόσο ενδιαφέρουσες ε, πληροφορίες. Ε, πρόκειται για αυτή την πρώτη εβδομάδα. Ήταν το ροντάρισμα, η δοκιμή. Αλλά είχαμε τέτοια συμμετοχή και επίσης ήταν σημαντικό το ότι είχαμε τις συνεργασίες για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Συνεργασία και με μη κερδοσκοπικές ε, ενώσεις και με τις ομοσπονδίες. Πολύ σημαντικός ο ρόλος τους όσον αφορά την πρόθεση του αθλητικού πνεύματος. Για πέστε μου, συναδελφοί, θέλετε να λάβετε το λόγο, κύριε Φίσα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας για να εκπροσωπήσω το Κοινοβούλιο, όπως είπατε, για την έναρξη της εβδομάδας των Βρυξελών. Ήταν μια επιτυχία σε συνεργασία με τον Επίτροπο, αλλά και τον Λουξεμβούργιο Υπουργό. Όλα πήγαν πολύ καλά. Όλα τα περίπτερα, τα στάντ, ε, τα διάφορα φιλικά γεγονότα και στην Μαδρίτη επίσης πήγα για την, τα εγγένεια της εκεί εβδομάδας και εκεί τα πήγαμε πολύ καλά. Οπότε πάμε, πήγαμε στο Σαν Σεμπαστιάν στη συνέχεια. Γιατί αυτή τη βδομάδα θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε επίσης και την ε, έκθεσή μας που υποστηρίζει τα παραδοσιακά αθλήματα, τα συλλογικά αθλήματα. Και στο Σαν Σεμπαστιάν αυτά θα προβληθούν, τα βασικά παραδοσιακά σπορ. Μα ξέρετε το Σαν Σεμπαστιάν επίσης είναι πολιτιστική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, οπότε θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ για αυτά τα παραδοσιακά σπορ. Και έτσι θα συμπέσει η εκδήλωση μία με την άλλη. Άλλωστε, τα σπορ είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και καλά κάνουμε εμείς και τα προωθούμε. Τα σπορ. Όπως σωστά είπε, είπε από την Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα είναι κάτι το οποίο το, το, το αναφέραμε στην έκθεση σαν η ημέρα αθλητισμού, η ημέρα έγινε εβδομάδα Οπότε στον Επίτροπο Επίτροπο να βράξει συγχαρητήρια αλλά και στον Επίτροπο Βασιλείου. Και η Επίτροπος ε, δεσμεύτηκε αυτή ότι θα ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το θέμα. Αλλά κύριε Λοστέκη θα σας πω ότι αυτή η εβδομάδα αθλητισμού δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι μια ευκαιρία να προβληθεί η σημασία του αθλητισμού στη ζωή μας. Και από κοινωνική σκοπιά έχουμε ένα σωρό ε, υπέρ, τα οποία ε, ε, είναι πάρα πολύ καλά για την υγεία, τα σπορ, βλέπουμε τόσα στοιχεία για τους νέους, για τους μεγαλύτερους, όπου ο αθλητισμός μπορεί μακροπρόθεσμα να ωφελήσει πάρα πολύ το κόστος των υπηρεσιών υγείας. Να, επομένως και μια άλλη έκθεση που λέγαμε για τη σχέση με την διατροφή, γιατί έχουμε την Αμερική πολύ ενσχετικά μέσα ότι αν κανείς δεν έχει διατροφή σωστή και αθλητική δραστηριότητα, τότε για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας μπορεί να έχουμε μία γενιά που θα έχει προσδόκιμο ζωής πιο κάτω από την προηγούμενη γενιά. Άρα να το πάρουν πολύ σοβαρά αυτό. Να, ο ρόλος του αθλητισμού. Οπότε και εγώ τώρα να σας πω κάτι, το ότι θα πρέπει να δούμε ότι είμαστε ενώπιον σημαντικού προβλήματος που είναι η μετανάστευση στην Ευρώπη. Ο καθένας έχει τις πολιτικές του απόψεις και για το θέμα αυτό, αλλά θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να έχουμε κάποια γηπεδάκια στα στρατόπεδα των προσφύγων. Απλά πράγματα. Και εκεί να μπορούν να κάνουν σπορ οι μικροί, οι μικρές, οι νέοι, οι νέες. Οπότε αυτό σας το ρίχνω έτσι σαν πρόταση και προς την Επιτροπή και προς τα κράτη-μέλη γιατί μπορούμε με λίγα χρήματα να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που τώρα είναι σε τόσο δύσκολη θέση. Πάντω και από οικονομική πλευρά ο ελληνισμός είναι πολύ σημαντικός, έμεσα άμεσα έχουμε αυτού που παράγουν το, το υλικό, τα φυσικά είδη, ε, τον τομέα των κατασκευών, από κάθε πλευρά. Είναι ηλικιώδη τα νούμερα, περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο κλάδο. Άρα και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επίσης, βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρον, θα συμφωνούν και οι συνάδελφοι, ότι του χρόνου θα έχουμε επίσης μία εβδομάδα αθλητισμού. Καλύτερα να μην συμπίπτει εβδομάδα του Στρασβούργου βέβαια, γιατί νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να συμμετάσχουμε περισσότερο. Όντα εδώ στις Βρυξέλλες θα ήταν καλύτερα. Εδώ βάζω τελεία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, έχετε δει και αυτό ήταν λίγο ανεπιτυχές ε, το ότι συνέπεσε με το Στρασβούργο. Θα πρέπει το χρόνο να το προσέξουμε αυτό. Νέκοφ και μετά λάβουν υπόψη τρεις ε, προσκεκλημένους. Κύριε Νέκοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα. Θα προσπαθήσω να είμαι συγκεκριμένος. Ως πρόσωπος της Κομισιόν για τη διπλή Όπως ξέρετε, πρέπει να σπουδάσουν ταυτόχρονα με την πραγματοποίηση της αθλητικής τους καριέρας. Και στο τέλος της αθλητικής σταδιοδραμίας πρέπει να αλλάξουν δουλειά. Να αλλάξουν δουλειά. Η Κομισιόν το κατάλαβε, το ένιωσε αυτό το πρόβλημα και το 12 δημοσίευσε μια ανακοίνωση γι' αυτό. Την ερωτώ λοιπόν παρακολουθείτε στενά τη συνέχεια που δόθηκε στο κείμενο εκείνο. Όσο για τον έρασμο, το πρόγραμμα έρασμος και το έρασμος συν η διπλή αυτή σταδιοδρομία είναι τμήμα του έρασμος συν και έχει και μεγαλύτερο πραϋπολογισμό για να αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα της διπλής σταδιοδρομίας και γενικότερα να αντιμετωπίσει το θέμα της απασχόλησης των νέων. Μετά το πρώτο έτος εφαρμογής του γνωρίζετε τι ποσοστό σχεδίων προγραμμάτων σχετίζονται και έχουν πραγματοποιηθεί για αυτή τη διπλή σταδιοδρομία. Ξέρουμε επίσης ότι ετοιμάζει η Κομισιόν κάτι για την ποιότητα των υπηρεσιών σε αυτές τις διπλές σταδιοδρομίες. Έχουμε τα ελάχιστα κριτήρια που χρειάζονται για να διασφαλίζεται η ποιότης. Ευχαριστώ. Ναι, αυτό αφορά ε, κάτι το οποίο αναφέρθηκε, αλλά αν μπορείτε κάνετε πιο συγκεκριμένες ερωτήσει. Βέντα. Σχετικά με τις παρουσιάσεις που ακούστηκαν και με την έκθεση ΦΥΣΑΣ, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη. Ε, παρακολούθησα πρόσφατα μια πολύ ενδιαφέρουσα τοπική αθλητική διοργάνωση στην ε, Ισπανία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, αλλά θα πρέπει να γίνεται ευρύτερα γνωστή. Πολύ συχνά υπάρχουν διάφορες ομάδες τη κοινωνία που έχουν την αίσθηση ότι δεν είναι προσβάσιμος ο αθλητισμός, ενώ στην πραγματικότητα είναι πάρα πάρα πολύ επωφελής ο αθλητισμός για όλε τι ηλικιακέ ομάδε. Ξέρω και από τη δική μου χώρα, όσον αφορά τα μικρά παιδιά, ηλικίας 6 έως 18 ετών ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για να ενθαρρυθούν νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και αν μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με ομάδες, με συλλόγους τα λοιπά. Αυτό είναι θετικό. Λοιπόν, έγινε η Ευρωπαϊκή Ομάδα Αθλητισμού. Στο μέλλον τι θα γίνει, ποιο είναι το επόμενο, το επόμενο διάστημα, τι θα γίνει. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο, πρέπει να ε, βρούμε συνεργάτες, πρέπει να βρούμε ανθρώπους, φορείς, οι οποίοι θα μπορέσουν να προωθηθούν, ε, να προωθήσουν τον, τον αθλητισμό. Και εγώ προέρχομαι από τον τομέα του, από τον του αθλητισμού και νομίζω ότι το Εράσμους Plus θα μπορούσε να προωθήσει ακόμη περισσότερο τον ε, αθλητισμό ώστε να έχουμε ακόμα θετικότερες επιπτώσεις στην κοινωνία. Μπορεί να μιλάει ένα ε, από τους αδέλφους και ένας ε, από τους προκεκλημένους των φορέων. Κίρκεμπι, πρόεδρος της ΣΥΣΚΑ, Διεθνής Φορέας Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχετε μια σημαντική εμπειρία από όλες τις ε, ομοσπονδίες και ξέρετε πώς μπορεί να προωθεί ο αθλητισμός από τη βάση της κοινωνίας. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να μιλήσω, να θέσω ερωτήματα, αλλά πολύ σύντομα. Η συμμετοχή είναι κάτι που γίνεται όλο και σημαντικό και για σένα David Walls, αλλά και για την Anna Kleisner. Αν δείτε τις δυνατότητες ανάπτυξης που υπάρχουν στον αθλητισμό, η οικονομική συμμετοχή ίσως είναι η σημαντικότερη. Η μεγαλύτερη συμμετοχή θα αυξήσει και τις οικονομικές επιπτώσεις. Δυστυχώς όμως υπάρχει και μια άλλη οικονομική επίπτωση από την αντίθετη πλευρά. Και αναφέρομαι στην απουσία φυσικής άσκησης. Εμείς απευθυνθήκαμε στον αρμόδιο επίτροπο και ρωτήσαμε αν μπορεί να βρει το κόστος της ε, απουσίας φυσικής άσκησης στην ε, Ευρώπη. Και μας απάντησαν ότι πρόκειται για 8 δισεκατομμύρια, 80 δισεκατομμύρια. 80 δισεκατομμύρια λοιπόν είναι το κόστος της απουσίας φυσικής άσκησης στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Επίσης η απουσία αυτή κοστίζει μισό εκατομμύριο ζωές κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Άρα, λαμβάνοντας υπόψη ποιο είναι ο συνολικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η παροχή και η εξασφάλιση της ειρήνης και της ευημερία στους λαούς της, έχουμε ηθική αλλά και οικονομική υποχρέωση να αυξήσουμε σημαντικά το επίπεδα φυσικής άσκηση. Ε, άσκησης. Είμαστε εταίρος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Αθλητισμού, την υποστηρίζουμε και ίσως εμείς ε, συμβάλαμε και στο να γίνει εβδομάδα και όχι ημέρα και εμείς υποστηρίζουμε την ε, διοργάνωση αυτή από τη σκοπιά του μαζικού ε, αθλητισμού. Εμείς έχουμε επίσης εκπονήσει και μια εκστρατεία με τον τίτλο Now We Move, τώρα κινούμαστε, μπορεί και να έχετε δει και τα υλικά μας και αυτό που ε, χρησιμοποιούμε ως εμβληματική διοργάνωση είναι η εβδομάδα κίνησης, μια ε, εβδομάδα που ε, πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο και μπορώ να σας πω κύριε Λοστέκ ότι μπορούμε να συνδέσουμε αυτές τις δύο διοργανώσεις την Ευρωπαϊκή Ομάδα Αθλητισμούς με το Move Week γιατί όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτές τις διοργανώσεις έχουν ένα στόχο, να σηκώσουν τους ανθρώπους από τον καναπέ τους. Έχουμε λοιπόν κάθε προθυμία να συμβάλλουμε και εμείς. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ομάδα Αθλητισμού είναι ένα θετικό βήμα και ελπίζουμε να υπάρξει περισσότερη προσοχή στον, στο, στο μέλλον στο να εξασφαλιστεί η ειρήνη και η ευημερία των ε, πολιτών της Ευρώπης. Ευχαριστούμε για αυτές τις προτάσεις. Η Τζούλι Βόρντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθώ και αυτή τη φορά. Έμαθα πολλά. Συνήθως αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι, η τέχνη και ο πολιτισμός, γιατί από εκεί προέρχομαι πριν, πριν ασχοληθώ με την ε, πολιτική και πολλές φορές υπάρχει αυτός ο, ο διαχωρισμός μεταξύ πολιτισμού και αθλητισμού και μ' αρέσει που εδώ στην Επιτροπή μας τα εξετάζουμε μαζί αυτά τα δύο, αυτούς τους δύο τομείς. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, το έργο σας κύριε Χένρι γιατί είμαι εισηγήτρια για την διαπολιτισμική μάθηση και τις θημελιώδες αξίες και η αλήθεια είναι ότι μα έλειπε αυτό το κομμάτι του αθλητισμού και αυτά τα στοιχεία που μα δώσατε σήμερα είναι πραγματικά ουσιώδη στοιχεία που, χρειαζόμαστε για την ε, σύνταξη αυτής της ε, έκθεσης. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε σήμερα εδώ και που διευκολύνατε το έργο μου ως εισηγήτρια στη σύνταξη της συγκεκριμένη έκθεσης. Είπαμε ένας από μια οργάνωση και ένας ε, συνάδελφος. Ε, Αλόνσο τώρα για κάποια ευρωπαϊκή συνοσπονδία αθλητισμού. Και κατόπιν θα λάβει το λόγο η κυρία Τρούπελ. Κυρία Πρόεδρε Κώστα, σα ευχαριστούμε συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία τη σημερινή για να λύσουμε τον αθλητισμό. Ευχαριστούμε και για την εβδομάδα και συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμμετάσχαμε ε, ως, ως φορέας των ε, ευρωπαϊκών πρωτευουσών για τον αθλητισμό. Είχαμε για ένα toolbox από διάφορους ε, φορείς. Όλοι αυτοί είναι όπως η ίσκα, όπως η φύση ε, βασικοί συνεργάτες για την εβδομάδα. Και εμείς ε, έχουμε αυτό το δίκτυο των ευρωπαϊκών πόλεων, συμμετέσχουν 18 πόλεις από 18 χώρες, είχαμε δραστηριότητες για τους ανήλικους στα σχολεία και άλλες δραστηριότητε την Κυριακή για τις οικογένειες αλλά και άλλες δραστηριότητε το Σεπτέμβριο ας πούμε στην Μποκλάβα στην Κροατία όπου 20% ε, του πληθυσμού συμμετέσχει πολύ σημαντικό το να εμπλακούν τόσοι άνθρωποι σε αθλητική δραστηριότητα Πάντως αυτό που θα πρέπει να γίνει, όπως έλεγε και ο συνάδελφος, είναι να μην μείνουν όλα αυτά στα πλαίσια μιας εβδομάδας αλλά αυτές οι δραστηριότητε να επικρατούν και στις 52 εβδομάδες του χρόνου. Το 2015 ε, το Τωρίνο θα έχει την, την Προεδρία όσον αφορά τα πολιτιστικά και εκεί έγινε μια συνάντηση, μιλήσαμε ε, για την εβδομάδα του αθλητισμού, για, τους, ε, για τις προκλήσεις που θα έχουν οι πόλεις στο μέλλον και όπως τα είπε και ο κύριος Φίσας είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να μετακινηθεί λίγο ε, σε άλλη εβδομάδα, εκτός Στρασβούργου η εβδομάδα της Ευρώπης, αλλά θα πρέπει όχι μόνο το Στρασβούργο να μην συμπέσει, αλλά να μην συμπέσει και με την έναρξη των ε, σχολείων για να συμμετάσχουν τα παιδιά. Κάτι άλλο τώρα, ε, εμείς από πλευράς των ευρωπαϊκών πρωτευουσών προτείνουμε του χρόνου την Πράγα, να είναι αυτή η πρωτεύουσα του αθλητισμού για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τίποτα άλλο ε, και επίση του χαιρετισμού από την πρόεδρο τη Οργανισμού είναι εδώ. Ευχαριστούμε και τώρα συνάδελφο Τρούπελ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους παρευρέθηκαν σήμερα εδώ στο πάνελ και θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στον κύριο Χένρι γιατί χάρηκα ιδιαίτερα με τα αποτελέσματα των μελετών και των ερευνών που αναφέρατε και φαίνεται ότι υπάρχουν θετικές επιπτώσεις του αθλητισμού σε ε, ομάδες προσφύγων και μεταναστών και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά το κοινωνικό κεφάλαιο στις κοινωνίες μας. Ε, γιατί γνωρίζετε αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες που έρχονται προς τη Γερμανία, τη Σουηδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και νομίζω ότι ιδιαίτερα οι αθλητικές δραστηριότητες για πολλούς από αυτούς τους πρόσφυγες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να μάθω αν ε, συμμερίζεστε εσείς αυτήν την άποψη ότι θα πρέπει να προσφέρονται περισσότερες δυνατότητες άθλησης σε αυτούς τους ε, πρόσφυγες που έρχονται ε, την περίοδο, περίοδο αυτή ε, στην Ευρώπη. Σίγουρα και συμφωνώ με αυτό το οποίο λέτε βεβαίω και ω Επιτροπή Πολιτισμού μπορούμε όλοι μαζί να προωθήσουμε αυτό που λέτε και τώρα να δώσουμε τον ε, λόγο στον κύριο ε, Μπίκη που είναι ο εκπρόσωπος τη ΦΙΖΗ που είναι εκπρόσωπος της βιομηχανίας αθλητικών ειδών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ Σιλβία για την ευκαιρία που μας δίνετε να ε, παρευρεθούμε εδώ. Συγχαρητήρια σε σένα, σε εσά και σε όσους διοργάνωσαν αυτό το workshop. Είμαι ο Αλμπέρτο Μπίκη, είμαι Γενικός Διευθυντής της ΦΙΖΗ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγής Αθλητικών Ειδών. Adidas, Nike, Puma, αυτά είναι τα μέλη μας. Εκπροσωπούμε 1.800 εταιρείες του κλάδου και συμβάλλουμε σημαντικότατα στα ε, αποτελέσματα που κατακτήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Αθλητισμού που επιτέχθηκαν. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο πτυχές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για μένα. Πρώτον, αυτό που κάναμε ως ε, ε, κλάδος για την Ευρωπαϊκή Ομάδα Αθλητισμού και δεύτερον θα ήθελα να αναφερθώ και να σας δώσω την δική μας πρώτη εικόνα για αυτή την, αυτή, για αυτή την Ευρωπαϊκή Ομάδα Αθλητισμού. Πρώτα απ' όλα να θέσουμε, προσπαθήσαμε να επηρεάσουμε και το περιεχόμενο αυτής της εβδομάδας αθλητισμού. Για παράδειγμα, ε, κοινοποιήσαμε ε, ερευνητικά πορίσματα ε, μιας έρευνας που είχαμε διοργανώσει πριν από κάποια χρόνια, το Design to Move. Αυτή ήταν η δική μας συμβολή από ερευνητικής άποψης είναι ε, σημαντικό να γνωρίζετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ε, εύρος στοιχείων και ανάλυσης που έγινε στο πλαίσιο αυτής της μελέτης. Το δεύτερο πράγμα που προσπαθήσαμε να κάνουμε όλα τα μέλη της ε, Ομοσπονδίας μας αλλά και οι ε, λιανικοί έμποροι και αναφέρθηκαν και αυτοί εμάς μας ενδιαφέρει βεβαίως ε, ιδιαίτερα η οικονομική επίπτωση του αθλητισμού, αλλά ε, προσφέραμε και μορφές επικοινωνίας. Ε, αναφέρθηκαν οι πρεσβευτές και συμβάλαμε και εμείς με παρέχοντας ναι, μεγάλα ονόματα όπως ο Steve Gerrard, η Paula Radcliffe αλλά και λιγότερο διάσημους αθλητές όπως η Gerlinde Kaltenbrunner, η οποία παρευρέθηκε και στην εναρκτήρια εκδήλωση μαζί με τον Σαντιαγό ε, όπως και ο Πίτροπος Ναβράσκης. Ε, επίσης υποστηρίξαμε με διάφορα δώρα αυτή την διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ομάδας ε, Εβδομάδας Αθλητισμού. Είμαστε συνδιοργανωτές της εκδήλωσης και ο τρίτος που βάλαμε είναι ο συντονισμός. Δημιουργήσαμε το επίσημο άνοιγμα μάλλον ε, της εκδήλωσης ήταν την ε, προηγούμενη Πέμπτη. Έχουμε, ε, είχαμε τα εγγένεια ενός, κριτή, ενός κτηρίου διαφόρων οργανώσεων και ομοσπονδιών με τέσσερις στόχους. Η οικονομική διάσταση, η, οικονομική, κοινωνική διάσταση, η διάσταση της υγείας, η διάσταση της αρκεραιότητας στον αθλητισμό. Είναι λίγο πολύ τα θέματα που ε, απασχόλησαν και τους ομιλητές της σημερινής εκδήλωσης και αυτό που θέλω να πω τέλος είναι η γνώμη μας για την Ευρωπαϊκή ε, Εβδομάδα Αθλητισμού. Υπάρχουν πάντοτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε ό,τι και αν κάνει κανείς βεβαίως. Αλλά οπότε θα, ε, θα σας πω ένα μεγάλο πλεονέκτημα και ένα μεγάλο ε, μειονέκτημα. Το πλεονέκτημα βεβαίως είναι το γεγονός ότι στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία η διοργάνωση. Λόγω των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν άνω των 3.000 ε, εκδηλώσεων λόγω του αριθμού των χωρών που συμμετείχαν σε αυτή την πρώτη Ευρωπαϊκή Ομάδα Αθλητισμού. Άρα είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και χαρούμενοι για την ε, ολοκλήρωση αυτής της πρώτης Ευρωπαϊκής Ομάδας Αθλητισμού. Φυσικά θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα και εδώ συμφωνώ με την άποψη του κυρίου Φίσας για το γεγονός ότι η επόμενη διοργάνωση της εβδομάδας του δεν θα πρέπει να συμπέσει με ολομέλεια στο Στρασβούργο. Και τέλος νομίζω ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ποιο είναι ε, το κοινό στόχος που έχουμε και ποιο θα είναι το μήνυμα που θα αποστέλλεται μέσα από αυτήν τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Αθλητισμού. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η σχετική μοίρα που διοργανώθηκε υπήρχε και υπουργική συμμετοχή, ήταν πολύ σημαντικά όλα αυτά, οι επαφές δηλαδή του Κοινοβουλίου με τους διάφορους φορείς. Ε, όπως γνωρίζετε εσείς που είστε εδώ, ε, μπορείτε να θέλετε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Έχω και εγώ κάτι να ρωτήσω για τον ε, άρμο της Επιτροπής και οι υπόλοιποι όμως μπορείτε να απαντήσετε, να μας πείτε σκέψεις σας. Μπορεί να αρχίσει Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περιοριστώ σε δύο-τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη για τον Σαντιάγο Φίσας. Ο παραδοσιακός και αθλητισμός της υπαίθρου είναι όντως κάτι σημαντικό και αυτή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού θέλουμε να τονίσουμε και τον παραδοσιακό αθλητισμό όπως το είχε ψηφίσει το 13 ήδη το Κοινοβούλιο και θα υπάρξει και συνέχεια γιατί το 16 στα πλαίσια του Εράσμου ΣΥΝ θα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών των παραδοσιακών μορφών αθλητισμού. Τώρα για τη διπλή σταδιοδρομία πράγματι θέλουμε να εφαρμοστούν οι συστάσεις βάζοντας προτεραιότητα στο έρασμος συν το 2014 είχαμε 14 εκατομμύρια στο πρόγραμμα συνεργασίας, εξών 7 στους δύο τομείς όπου υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές. Εξών και η διπλή σταδιοδρομία. 3,5 εκατομμύρια για το Joel Carrier. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξαν πολλές αιτήσει και χρηματοδοτήσαμε μόνο δύο προγράμματα, ένα εκατομμύριο επί 3,5 εκατομμυρίων δηλαδή μόνο ένα μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε. Το 2015 το ξαναζητήσαμε και θα δούμε σε δυο 3 εβδομάδες τι σχέδια θα έχουν υποβληθεί. Πράγματι πάντως η Κομισιόν θέλει να εφαρμοστούν οι συστάσεις για τη διπλή σταδιοδρομία. Τέλος, και να απαντήσω στον κύριο Βέντα, για τη συνέχεια είναι πράγματι ουσιώδες όχι μόνο κατά την εβδομάδα εορτασμού αλλά και τις υπόλοιπες. Οι εταίροι μας έχουν όλοι αναλάβει ευθύνες μακροπρόθεσμα, όχι μόνο μερικές δραστηριότητες μία εβδομάδα. Δεύτερον, στις οικονομικές εταιρικές σχέσεις που έχουμε συνάψει, δεν πρόκειται μόνο για δεκαπενθήμερα προγράμματα αλλά πιο μακροχρόνια. Ας σταματήσω εδώ και ευχαριστώ όλους τους εταίρους μας που είναι εδώ στην αίθουσα όπως το Φερσίτο, Ατσές, Ίσκα και άλλους. Θέλει κάποιο άλλος να βέβαια τον λόγο για να κλείσει. Ε, σας ευχαριστώ όλους για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είδαμε σήμερα σε βάθος αυτά όλα ε, τα πρότυπα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τόσο ώστε να μπορέσει το σπορ να είναι παράγον συμπερίληψης, ένταξης, προσέγγισης. Julie Ward Έχουμε και τη δική σου έκθεση που είναι πολύ σημαντική όσον αφορά ε, την παιδεία που έχει το τόσα κοινά με την γιατί έχουμε τώρα και την οικονομική άποψη του αθλητισμού γιατί βλέπουμε ε, ότι θα έπρεπε στα πλαίσια ε, της αποτίμησης αυτής να έχουμε και τα αποτελέσματα της απουσίας της αθλητικής δραστηριότητα. γιατί υπάρχει κόστος από πλευράς ανθρώπινης από πλευράς δαπανών υγείας Υπάρχουν πολλές ε, δυσμενείς συνέπειες για την κοινωνία όταν υπάρχει σπορ. Υπάρχουν πολλά που μπορεί κανείς να εμβαθύνει εδώ. Τώρα δεν θα πρέπει όμως να ξεχνούμε και αυτά που είπε ο κύριος Βόλς ε, ε, που μας κατέθεσε την προσωπική του εμπειρία αυτά τα οποία λέγαμε και με τον κύριο Υπουργό δηλαδή για αυτές τις συμπεριφορές που δηλητηριάζουν τον αθλητισμό. Αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει με συγκεκριμένο τρόπο να ε, θεσπίσει κάποια νομοθετικά κείμενα για να αντιμετωπιστεί το ντόπινγκ. Αλλά, όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να θεσπίσει μια οδηγία και να γίνει αυτό το οποίο έχουν κάνει κάποιες χώρες. Για όλες τι χώρε δηλαδή, να ποινικοποιηθεί το ντόπινγκ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε επίση για όσου από εσά δώσατε τι ομιλίε σε όλου ανθρώπου για να ενημερωθούν. Οπότε εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ακρόασή μα. Και θα συνεχίσουμε με τη συνάντηση των συντονιστών. Και κλεισμένο των θυρών. Ευχαριστούμε και πάλι